So, uh, ladies, uh, ladies and gentlemen, dear, dear colleagues, uh, we have. Ladies and gentlemen, dear colleagues, we have a very. Αγαπητοί συνάδελφοι, έχουμε σήμερα μία μεγάλη ημερήσια διάταξη. Ως εκ τούτου πρέπει να προσπαθήσουμε να ξεκινήσουμε στην ώρα μας ακόμα και αν δεν είναι όλοι παρόντες. Θα ήθελα λοιπόν να σας ανακοινώσω ότι έχουμε τις ε, γλώσσες που αναφέρονται στα έγγραφα. Ε, οι άλλες ε, που δεν αναφέρονται, δεν, σε αυτές δεν υπάρχει διερμηνία. Έχετε λοιπόν μπροστά σας την ημερήσια διάταξη και αν δεν υπάρχουν παρατηρήσεις, εγκρίνεται η ημερήσια διάταξη. Τώρα πρέπει να επιλέξουμε κάτι. Συγκεκριμένα ο κύριος Σλότια, ο οποίος είναι ο τρίτος αντιπρόεδρος, ε, παρετήθηκε από τη θέση του Ευρωβουλευτή και το ΕΛΚ μπορεί να προτείνει τον κύριο Αμπράτσαν, τον οποίο και προτείνει τον αντικαθιστά. Αν λοιπόν δεν υπάρχουν αντιρρήσεις, ε, προτείνω ως τρίτο αντιπρόεδρο να έχουμε τον κύριο Αμπράτσαν ε, και να τον εκλέξουμε διαβοής. Ε, δεν ξέρω, βέβαια πρέπει καταρχήν να ρωτήσω, υπάρχουν άλλοι υποψήφοι, από ό,τι βλέπω όχι. Ως εκ τούτου συμφωνείτε και με τη διαδικασία και θα ε, πρότεινα η εκλογή να γίνει δια χειροκροτημάτων, δια Ε, σαφή τα χειροκροτήματα και ε, θα ήθελα λοιπόν να συγχαρώ τον νέο μας αντιπρόεδρο. Τώρα θα ήθελα να σας ε, υπενθυμίσω ότι έχουμε προβλέψει και μία επίσκεψη στον Ευρωπαϊκό Αμυντικό Οργανισμό την 5η 19 ε, Μαρτίου στις 9.30 ώρα το πρωί για δύο περίπου ώρες. Η επίσκεψη αυτή θα λάβει χώρα στις Βρυξέλλες και θα χαιρόμουν πολύ αν ε, στην επίσκεψη αυτή η παρουσία σας ήταν έντονη γιατί νομίζω ότι η συνεργασία ανάμεσα στη δική μας την Υποεπιτροπή και τον Αμυντικό Οργανισμό ήταν ε, ιδιαίτερα αγαστή και θα πρέπει να συνεχιστεί. Κατά τα άλλα στις 30 ε, Μαρτίου θα έχουμε την τελευταία μας συνεδρίαση για αυτή τη θητεία του Κοινοβουλίου και θα ήθελα να σας πω ότι στο τέλος της συνεδρίασης θα έχουμε και ένα εργαστήριο σχετικά με τις ε, στρατιωτικές εγκαταστάσεις των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τον ρόλο τους για την ΚΕΠΑ. Προβλέπετε η διεξαγωγή αυτού του εργαστηρίου, workshop. Όπως επίσης πολλοί από εσάς ε, γνωρίζετε, εγώ δεν θα είμαι στο επόμενο Κοινοβούλιο Ευρωβουλευτής. Είναι η τελευταία μου θητεία. Γι' αυτό ε, όταν θα έχουμε την τελευταία μας συνεδρίαση στις 30 Μαρτίου, μετά στο τέλος θα ήθελα να σας ε, καλέσω σε μία μικρή δεξίωση για ποτό. Σήμερα λοιπόν έχουμε τη χαρά να ε, μπορούμε να καλωσορίσουμε την κυρία Κατερίνα ε, Σεκουάνισοβα ε, η οποία θα μας ενημερώσει αλλά τηλεγραφικά θα ήθελα να πω ότι η εφαρμογή του κώδικα συμπεριφορά για τι εξαγωγέ όπλων ε, μέσω μια κοινή θέση είναι κάτι το ευπρόσδεκτο για όλου μα. Κατά τη διάρκεια αυτή τη ε, κοινοβουλευτική θητεία, ένα ε, στόχο τη υποπιτροπή μα ήταν ακριβώ αυτό, να επιτύχουμε κοινή θέση και αυτός ο κώδικας ε, συμπεριφοράς να καταστεί δεσμευτικός σε όλα τα κράτη-μέλη. Χαιρετίζω λοιπόν ιδιαίτερο το γεγονός ότι το επιτύχαμε αυτό. Και κατά δεύτερον θα ήθελα επίσης ε, να πω ότι ε, στην Armstrong.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 του ΣΚΟΑΡΜ με τον πρόεδρο και τα μέλη της υποεπιτροπής σας. Ο κύριος Jean-Claude ο προκάτοχός μου, σας ενημέρωσε στις 8 Δεκεμβρίου του 2008 ε, και είναι τιμή για μένα που βρίσκομαι εγώ εδώ σήμερα. Έχω έρθει βέβαια νωρίτερα κατά τη διάρκεια του εξαμήνου για προφανείς λόγους. Και αυτός είναι και ο λόγος γιατί θα ήθελα να σας ε, παρουσιάσω τις ε, πληροφορίες μου κατά θέματα και όχι κατά χρονολογική σειρά. Πρώτα απ' όλα θα ήθελα να σας αναφέρω κάποιες λεπτομέρειες σχετικά με την έγκριση και την εφαρμογή της ε, κοινή θέσης 944 της 8 Δεκεμβρίου του 2008 όπου αναφέρονται κοινοί κανόνες που θα διέπουν την εξαγωγή ε, στρατιωτικού εξοπλισμού και στρατιωτικής τεχνολογίας. Δηλαδή με άλλα λόγια την θέσπιση του κώδικα συμπεριφοράς ως κοινή θέση. Η κοινή θέση είναι ένα νομικά δεσμευτικό έγγραφο το οποίο αντικαθιστά τον πολιτικά δεσμευτικό κώδικα για, την, ε, για το εμπόριο όπλων. Προβλέπει ότι τα κράτη-μέλη ε, πρέπει να αξιολογούν τις άδειε για την εξαγωγή όπλων σύμφωνα με τα κριτήρια που αναφέρονται στο άρθρο 2. Πιο συγκεκριμένα το, τα κριτήρια ε, που συμπεριλαμβάνονται στο άρθρο 2 μοιάζουν με εκείνα τα οποία ε, γνωρίζετε από τον κώδικα συμπεριφοράς. Παρόλα αυτά υπάρχουν κάποιες ε, διαφορές, η κοινή θέση διευρύνει το στόχο του αρχικού κώδικα συμπεριφοράς. Κυρίως θα ήθελα να σας επισημάνω ότι μία από τις μικρές διαφορές που υπάρχει ε, ανάμεσα στον κώδικα συμπεριφοράς και την κοινή θέση είναι το κριτήριο υπαριθμών 2 το οποίο περιλαμβάνει σαφή αναφορά στο διεθνές ανθρωπιστικό δίκαιο κάτι το οποίο δεν συνέβαινε στον κώδικα συμπεριφοράς. Έτσι λοιπόν η ΚΟΑΡΜ ε, σύντομα ε, θα σας παρουσιάσει μια επικαιροποιημένη εκδοχή του εγχειριδίου Χριστών θα διαπιστώσετε ότι αυτό είναι ένα έγγραφο ε, δημόσιο το οποίο το συνέταξε η ΚΟΑΡΜ και ε, παρουσιάζει λεπτομέρειες για τον κώδικα συμπεριφοράς και την κοινή θέση και πώς αυτά τα δύο πρέπει να ερμηνεύονται. Επίσης ε, τα κράτη-μέλη κάνουν τα απαραίτητα βήματα για να διασφαλίσουν ότι θα υπάρχει ειδική αναφορά στην κοινή θέση και τούτο μάλιστα στην εθνική τους νομοθεσία. Οι τρίτες χώρες οι οποίες είχαν υιοθετήσει τον κώδικα συμπεριφοράς μας ενημέρωσαν ήδη ότι είναι πρόθυμες να προσαρμοστούν στην κοινή θέση. Όσον αφορά τώρα στην έγκριση του κώδικα συμπεριφοράς ως ένα δεσμευτικό νομικό έγγραφο, αυτό είναι ένα σημαντικό μήνυμα προς την κοινή γνώμη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και γενικότερα προς ολόκληρο τον κόσμο, ότι δεν θα πρέπει να εξάγονται όπλα ε, τα οποία θα χρησιμοποιούνται για καταπίεση, για επιθετικότητα ή που θα συμβάλλουν στην περιφερειακή αστάθεια. Η νομικά δεσμευτική κοινή θέση επίσης αποτελεί ένα παράδειγμα για τη συνεργασία των συστημάτων ελέγχου και ενισχύει την αξιοπιστία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αποδεικνύει το εφικτό ε, των, ε, της Διεθνούς Σύμβασης ε, περί εμπορίου όπλων και φτάνω λοιπόν τώρα στο επόμενο θέμα το οποίο είναι πρώτη προτεραιότητα για την τσεχική προεδρία όσον αφορά τις αρμοδιότητες της ΚΟΑΡΜ. Στόχος μας είναι να προάγουμε τη διαδικασία που θα οδηγήσει στην έγκριση της συνθήκης της ATT. Όπως πολύ καλά γνωρίζετε, η Ευρωπαϊκή Ένωση στο σύνολό της, αλλά και τα μεμονωμένα κράτη-μέλη υποστηρίζουν αυτή την συνθήκη που έπεται και εδώ παίζει ρόλο το ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου του Ιουνίου του 2007. Όλα τα κράτη-μέλη προτίθενται να συνεχίσουν να διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο στη στήριξη αυτού του στόχου. Με την ιδιότητά μου ως Προέδρου της COARM εγώ να από κάποιες εβδομάδες συμμετείχα στην ε, πρώτη ομάδα εργασίας ε, χωρίς καταληκτική ημερομηνία που συνεκλήθη στη Νέα Υόρκη και με χαρά μου μπορώ να σας ε, πω ότι τα αποτελέσματα αυτής της πρώτης συνάντησης είναι θα έλεγα, θα τα χαρακτήριζα ενθαρρυντικά. Υπήρξε μια συνάντηση οργανωτικής φύσεως τον Ιανουάριο που δεν ήταν όμως τόσο ενθαρρυντική, ασχολήθηκε περισσότερο με οργανωτικής φύσεως ίσως θέματα και μεθόδους εργασίας. Όμως ε, ευτυχώς ε, χάρη ε, τον, του πρέσβη Μοριτάν, του ικανότατου πρόεδρου, ο οποίος προείσταται αυτή τη ομάδα εργασία στη Νέα Υόρκη, συμφωνήθηκε ήδη την πρώτη μέρα η μερίσια διάταξη, που σημαίνει ότι κατά το υπόλοιπο αυτή τη εβδομάδα μπορέσαμε να συζητήσουμε την ουσία του θέματος και να επικεντρωθούμε σε στόχους, σε ε, παραμέτρους μιας ε, επικείμενης ε, συμφωνίας, συμφωνίας ATT. Κατά τη διάρκεια λοιπόν αυτών των συζητήσεων κατέστη σαφές ότι τα κράτη-μέλη χωρίζονται σε τρεις κατηγορίες. Η πρώτη αφορά τους αμύντορες. Εδώ Έχουμε ε, χώρες Ευρωπαϊκής Ένωσης ε, και άλλες ε, χώρες με ίδιες απόψεις εκτός των Πολιτειών. Οι χώρες υποσαχάριας Αφρικής, Λατινική Αμερική ή αν θέλετε Ινδονησία και κατόπιν έχουμε στη δεύτερη κατηγορία τις επιφυλακτικές χώρες που είναι Ρωσία, Κίνα, Ινδία, Ισραήλ και οι περισσότερες αραβικές χώρες και κατόπιν τρίτη κατηγορία οι αντίθετες χώρες Πακιστάν και Αίγυπτος. οι Ηνωμένε Πολιτείε αποτελούν ε, κατηγορία αυτή καθεαυτή που όπως γνωρίζετε καταψήφισαν ε, το ψήφισμα που προέβλεπε τη σύσταση αυτής της ομάδας εργασίας χωρίς καταλακτική ημερομηνία η οποία πρόκειται να ασχοληθεί με τη συνθήκη. Με την αλλαγή βέβαια της κυβέρνησης η θέση των Ηνωμένων Πολιτείων δεν έχει ακόμα διευκρινιστεί και θα έλεγα ότι υπάρχει ακόμα περιθώριο για συγκρατημένη αισιοδοξία. Ιδιαίτερα συγκρατημένη αισιοδοξία. Εξάλλου, αυτό που κατέστησε σαφέ κατά τη διάρκεια τη εβδομάδα αυτή στη, Νέα Υόρκη ήταν ότι δεν γνωρίζουν όλα τα κράτη-μέλη τι επιπτώσει και το λογικό που διέπει την επικείμενη συνθήκη. Ε, αυτό ισχύει κυρίως για εκείνες τις χώρες οι οποίες ε, δεν ε, εκπροσωπήθηκαν το 2008 με τη μορφή του κυβερνητικού εμπειρογνώμονα. Θα ξέρετε ότι το 2008 συναισθήθη μια ειδική ομάδα κυβερνητικών εμπειρογνωμών, 27 που συναντήθηκαν τρεις φορές και συζήτησαν για, την, για το εφικτό και τις παραμέτρους της συνθήκης, της ATT. Εφέτος άλλαξε λιγάκι η διάταξη αυτή, προχωρήσαμε περισσότερο. Είχαμε μόνο δύο συναντήσεις, αλλά με τη μορφή μιας ε, ε, ομάδας εργασίας ανοιχτή ημερομηνία, που δεν σημαίνει ότι οι συζητήσεις θα συνεχιστούν στο διηνεκές, αλλά ε, στην ομάδα αυτή μπορούν να συμμετέχουν όλα τα κράτη-μέλη που επιθυμούν. Έχοντας λοιπόν κατά νου την προαγωγή της συνθήκης ATT μπορώ να σε ενημερώσω ότι στις 18 Ιανουαρίου το Συμβούλιο ε, ενέκρινε την ε, έλαβε την απόφαση τη 42, παριθμό 42, έτσι ώστε να ε, προχθεί στις υποψήφιες χώρες η διαδικασία εκείνη που θα οδηγήσει στη συμφωνία ATT, Arms Trade Treaty, συμφωνία για το εμπόριο των όπλων. Η διαδικασία ξεκίνησε στη Γενέβη με μια εναρκτήρια τελετή, μια εβδομάδα πριν από την έναρξη εργασιών της ομάδας εργασίας και ο στόχος ε, ήταν να υπάρξει ενημέρωση των μόνιμων επιτροπών, των ε, εκπροσώπων, των ε, πρέσβεων για αυτές τις δραστηριότητες και για το γεγονός ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση διεξάγει ένα είδος προγράμματος προαγωγής, ενίσχυσης, στήριξης μάλλον της ATT. Η Αλίσα Τζανέλα και εγώ με την ε, ιδιότητά μας των ε, συμπροέδρων. Ήμασταν και οι δύο παρούσες κατά την εναρκτήρια τελετή και απευθυνθήκαμε στο φόρουμ με εισαγωγικές ομιλίες. τώρα, όσον αφορά την ουσία του ε, προγράμματος, προβλέπεται να λάβουν χώρα έξι περιφερειακά σεμινάρια, δύο για την Αφρική, ένα για τη Μέση Ανατολή, ένα για τη Λατινική Αμερική και την ε, Καραϊβική, ένα για την Ασία και τον Ειρηνικό και ένα για τις ε, χώρες του ΩΣΑ. Αυτά θα λάβουν χώρα στην Ευρώπη. Επίσης ε, προβλέπονται και άλλες συναφείς εκδηλώσεις. Μία εκδήλωση στο περιθώριο της πρώτης συνάντησης των Επιτροπών στη Νέα Υόρκη τον Οκτώβριο αυτού του έτους. Κατόπιν θα υπάρξει και απλά ε, σύντομα θα ήθελα να σας υπενθυμίσω ορισμένους στόχους όπως αυτό, αυτοί ακριβώς αναφέρονται στην απόφαση του Συμβουλίου. Υπάρχει, ε, υπάρχουν λοιπόν τα κράτη-μέλη των Εθνών, οι κοινωνίες των πολιτιών και οι βιομηχανικοί κύκλοι οι οποίοι συμμετέχουν στις συζητήσεις ε, για μια συμφωνία που θα συμβάλλει στην καλύτερη εμπλοκή των ΗΠΑ και των περιφερειακών οργανώσεων σε αυτή τη διαδικασία. Ανταλλαγή απόψεων ε, και προαγωγή των συζητήσεων ανάμεσα στα κράτη-μέλη, τις περιφερειακές οργανώσεις, τις κοινωνίες των πολιτιών και τη βιομηχανία. Επίσης ε, αξιολογήθηκαν επιπτώσεις από το ενδεχόμενο σύναψης μιας συμφωνίας ATT. Για να ανακεφαλώσω, ο στόχος είναι να υπάρξουν σε βάθος συζητήσει, να κινητοποιηθούν όλοι οι σημαντικοί παράγοντες και εδώ προφανώς θέλουμε να, ε, να ε, αποτανθούμε κυρίως σε όσους είναι επιφυλακτικοί. Η Γραμματεία του Συμβουλίου, η Προεδρία και τα κράτη-μέλη θα καταβάλουν κάθε δυνατή προσπάθεια για να διασφαλίσουν την, ε, το αίσιο τέλος, την επιτυχή κατάληξη αυτής της διαδικασίας ATT. Τώρα θα ήθελα να πω λίγα λόγια για τις δραστηριότητες της ΚΟΑΡΜΑ κατά τη διάρκεια της Τσεχικής Προεδρίας. Και Αυτές περιλαμβάνουν δραστηριότητες όσον αφορά, όπως ήδη είπαμε, το, την κοινή θέση για τον κώδικα διοντολογίας προφανώς. Επίσης ένα περιφερειακό σεμινάριο. Όπως ξέρετε υπάρχει μια κοινή δράση που βασίζεται σε ένα διετές πρόγραμμα και καλύπτει και θα, θα οργανωθούν διάφορα περιφερειακά σεμινάρια κατά την Γαλλική Προεδρία το περιφερειακό σεμινάριο το Σεπτέμβριο του 2008 είχε γίνει στο Ραμπάτ και εκεί είχαμε ε, συζητήσεις με 20 εκπροσώπους χωρών της Βόρειας Αφροκής και επίσης με στελέχη των Υπουργείων, των Άμυνας Τα Υπουργεία αυτά είναι υπεύθυνα για τη διοργάνωση παρομοίων σεμιναρίων στη Βόρεια Αφρική και με την εξαίρεση της Αιγύπτου όλες οι άλλες χώρες της Βόρειας Αφρικής ήταν παρούσες. Οι αντιπροσωπείες εστάλησαν από τις πρωτεύουσες των χωρών αυτών και στη, εκ μέρους της Λιβύης συμμετείχε και ένας εκπρόσωπος από τη Νέα Υόρκη. Όλη αυτή η συνεργασία γίνεται στα πλαίσια ε, της ε, συνεργασίας ε, καλής γυπνίασης της Ευρωπαϊκής Ένωσης με στόχο την συνθήκη ATT. Είπαν βεβαίως λέξη ότι όλοι είναι εναντίον της παράνομης εμπορίας ε, όπλων και ότι θα πρέπει να γίνει ένας αυστηρός έλεγχος κατά τη μεταφορά όπλων που βρίσκονται σε τράνζιτ διασυνοριακών μεταφορών και θα πρέπει επίσης να ελεγχθεί η μεταφορά όπλων για να μην διαταραχθεί η συνθήκη για τα συμβατικά όπλα και οι ήδη υπάρχουσες διεθνείς συμφωνίες. Υπό την ομπρέλα αυτή λοιπόν της κοινή δράσης κατά την Τσεχική Προεδρία θα γίνει μια περιφερειακή ε, συνεδρίαση στο Κίεβο, ε, Ουκρανία και εκεί θα συζητηθεί η συμμετοχή σε επίπεδο ευρωπαϊκό της Ουκρανίας σε ό,τι αφορά ακριβώς τον έλεγχο της ε, εξαγωγής όπλων. Το δεύτερο περιφερειακό σεμινάριο θα γίνει στα Δυτικά Βαλκάνια στα τύρανα και ε, ε, ανήκε στο πλαίσιο της συνεχούς προσπάθειας για τη συνέχιση των συζητήσεων μετά από τη Σλοβενική Προεδρία το Μάιο πέρσι, που είχε γίνει πέρσι το Μάιο. Το τελικό σεμινάριο λοιπόν σε αυτή τη διαδικασία της ε, κοινή δράσης θα γίνει υπό τη Σουηδική Προεδρία και θα καλύπτει τις χώρες Αρμενία, Ζερβαϊτζάν, Λευκορωσία και Μολδαβία. Και ε, υπό το φως της επερχόμενης ειδικής Προεδρίας και με την εμπειρία που έχουμε από τα τρέχοντα σεμινάρια θα πρέπει να αρχίσουμε να σκεφτόμαστε την ανανέωση της κοινή αυτής δράσης ε, αυτού του φορέα και ποιες χώρες θέλουμε να καλυφθούν στο μέλλον. Οι άλλες τρεις προτεραιότητες πέραν αυτών που ανέφερα είναι λοιπόν κοινή θέση για τον κώδικα διολογίας, η συνθήκη για τον έλεγχο εμπορίας όπλων, ATT και τα περιφερειακά σεμινάρια. Στις 13 Ιανουαρίου έγινε μια άτυπη συζήτηση στην Πράγα και όπως ξέρετε γίνονται τρεις επίσημες, τρεις επίσημες ε, συναντήσεις ε, αλλά το, στην αρχή κάθε Προεδρία ξεκινάει με τη διοργάνωση ενός άτυπου σεμιναρίου στην πρωτεύουσα και αυτό ήταν στις 13 Ιανουαρίου στην Πράχα. Ε, άλλες προτεραιότητες είναι ο συνεχής διάλογος με τους ε, εταίρους μας, δηλαδή με εσάς, τα μέλη της Ευρωπαϊκής, ε, του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και της Υποεπιτροπής Άμυνας και με πολλούς άλλους οργανισμούς. Επίσης θα ε, συνεχίσουμε την παράδοση προκαταρτικών ε, συναντήσεων με μη κυβερνητικού οργανισμούς. Κατά το τέλος Ιουνίου θα γίνουν αυτές οι συναντήσεις και θα συνεχίσουμε την κλασική παράδοση της, ε, των συναντήσεων Τρόικα ε, και τη συνεργασία με την Ρωσία και την Ορβηγία και τις Ηνωμένε Πολιτείε, ιδίω με τις Ηνωμένε Πολιτείε και τη Ρωσία είναι παρουσίαση ιδιαίτερα ενδιαφέρον η συζήτηση ε, στα, του πλαισίου της συνθήκης ATT. Είχαμε στο παρελθόν πολύ φιλικές συζητήσεις και δεδομένου ότι η Νορβηγία συμμετέχει στις συζητήσεις για τον κώδικα δεοντολογίας μέσα στην κοινή δράση, ανταλλάσσουμε υπόψεις κάθε τρεις μήνες τακτικά για να, για να υπάρξει αλληλό ενημέρωση. Η Τρόικα, η Καναδά, με Καναδά και Ουκρανία θα γίνει στο Μάιο βάσει της, ε, των ρυθμίσεων Βάσεμαρ θα ήθελα να πω ότι οι ρυθμίσεις Βάσεμαρ, ε, Βάσεναρ είναι άλλη μια διαδικασία την οποία θα συνεχίσουμε για να εξασφαλίσουμε και θέλουμε να εξασφαλίσουμε και τη συμμετοχή της Κύπρου σε αυτή τη ρύθμιση Βάσεναρ για να εξασφαλίσουμε ότι όλα τα μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι, είναι μέλη σε, αυτή την, σε αυτό το βασενάρ Arrangement. Τώρα, άλλα θέματα στην ημερήσια διάταξη είναι η διαδικασία υποβολής αναφορών, η, διαφάνεια, η έκθεση Σολάνα η οποία θα αναφέρει τις διάφορες άδειες που γίνονται εξαγωγής όπλων, πόσες υποβλήθηκαν, πόσες ε, δεν, εγκρίθηκαν, απορρίφθηκαν. Και η έκθεση αυτή θα συμπεριλαμβάνει και όλα τα συναφή στοιχεία από τα κράτη-μέλη. Θα κάνουμε επίσης μία ενημέρωση της, ε, ε, της έκθεσης ιδιωτικών στοιχείων και δεδομένων. Η τελευταία ολοκληρώθηκε το Δεκέμβριο και η ενημερωμένη έκδοση θα δημοσιευτεί στην επίσημη εφημερίδα της, ε, της Ευρωπαϊκής Ένωσης τέλος αυτής της εβδομάδος. Θα ήθελα επίσης να αναφέρω ότι παρακολουθούμε στενά και τη συζητή στο Συμβόλιο και στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για την κοινή οδηγία απλούστευσης των όρων και των κανονισμών για τη μεταφορά ε, ε, αμυντικού υλικού και συναφών ε, προϊόντων τα κράτη-μέλη ήδη μελετούν πώς είναι δυνατόν να μεταφερθεί στα εθνικά δίκαια με τον καλύτερο τρόπο η οδηγία αυτή όταν υιοθετηθεί. Είναι ένα άλλο σημείο αυτό σημαντικό στην ημερήσια διάταξη του μέλλοντος και με αυτά κύριε Πρόεδρε ολοκλήρωσα την παρουσίασή μου. Ευχαριστώ πολύ. Θα ήθελα να δώσω το λόγο τώρα στον κύριο Φλούγκα. Ευχαριστώ. Θα ήθελα κύριε Φονβόγκα να σας ακούσω πιο ενθουσιώδη διότι επιτέλους εδώ συζητάμε τον κώδικα δεοντολογίας μετά από τόσο καιρό. Έχουμε πραγματικά κουραστεί, έχουμε εργαστεί τόσο καιρό για αυτή την κοινή θέση και χαίρομαι ιδιαίτερα που καταλήξαμε σε αυτό το αποτέλεσμα. Άρα λοιπόν θα πρέπει να, έχουμε, ε, να είμαστε πανευτυχείς και ενθουσιώδεις. Ναι, ναι, καλά λέει ο πρόεδρος. Είμαι πρόθυμος να δείξω περισσότερο ενθουσιασμό. Απλώς είναι ο τρόπος μου έτσι. Ε, είμαι λίγο συγκρατημένος. Ίσως δεν δείχνω τόσο πολύ τον ενθουσιασμό μου. Δεν πειράζει, δεν πειράζει. Έχει καλός. Λοιπόν, τώρα τα προβλήματα στη μεταφορά της ε, οδηγίας ή της κοινής Τα, τα, τα πρακτικά προβλήματα. Θα ήθελα λοιπόν δύο ερωτήματα να θέσω για την πρακτική εφαρμογή. Ε, δεν ξέρω αν αυτό μπορεί να γίνει ε, συντάσσοντας μία έκθεση για τις συνέπειες και τις επιπτώσεις αυτού του κώδικα δεοντολογίας. Τα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης έχουν διεξαγάγει πολέμους, πολέμους ε, και έχουν συμμετάχει, έχουν αντιμετωπίσει πολέμους, παραδείγματο χάρη στη Γεωργία και στη Γάζα, στη Λωρίδα της Γάζας τι θα γίνει τώρα με τον κώδικα δεοντολογίας σε τέτοιες περιπτώσεις που θα παρουσιαστούν ή θα, προκύψουν οι πόλεμοι στο μέλλον. Θα πρέπει να ξέρουμε ακριβώς πώς και ποιος, ποιος παραδίδει και πώς γίνεται η παράδοση των όπλων. Διότι διαπιστώσαμε βεβαίως ότι χρησιμοποιήθηκαν όπλα και θα πρέπει να ελέγξουμε με μεγάλη προσοχή από πού την πηγή δηλαδή τον τρόπο μεταφοράς και τη χρήση των όπλων αυτών. Σε περιοχές κρίσεων και πολέμων οι εξαγωγές όπλων δεν θα πρέπει να επιτρέπονται πλέον. Δεν θα πρέπει να είναι δυνατόν να γίνονται ναι, είμαστε πολύ ευτυχείς με αυτή την εξέλιξη και θα ήθελα να ευχαριστήσω θερμά τη Γαλλική Προεδρία που εργάστηκε προς αυτό το στόχο και συνέβαλε στην εξέλιξη στην, αυτού του κώδικα δεοντολογίας μέσα στο, στο πλαίσιο της κοινή απόφασης έτσι ώστε να γίνει δεσμευτική. Πολλά χρόνια στο σώμα αυτό επιδιώκαμε αυτό το στόχο και είναι σημαντικό να τονίσουμε ότι η Γαλλική Προεδρία επέφερε αυτή την αλλαγή και έδωσε τη δυνατότητα πραγματοποίησης διότι πολλοί από εμά και εγώ είχα θέση τον δάκτυλο επί τον τύπων των είχα μάλλον ε, ε, κατηγορήσει τη γαλλική πλευρά ε, ότι παρακόλλησε ή κολυσιεργούσε και καθαστερούσε την, ε, το στόχο αυτόν, αλλά τώρα πρέπει να του συγχαρώ. δεν ε, είναι μόνο η Λευκή Βίβλος την οποία εξέδωσε η, Γαλλική Προεδρία πριν αρχίσει το, η, Γαλλική Προεδρία και δεν είναι μόνο ότι άλλαξε η νοοτροπία τους και η αντίληψή τους, διότι όπως ε, ξέρετε στη λευκή, η λευκή αυτή βίβλος δεν παρουσιάζει καμία αλλαγή. Λέει ότι περίπου ότι το status quo θα ισχύσει και όλα είναι ωραία και καλά και θα συνεχιστούν όπως ήταν. Τώρα λοιπόν βλέπετε ότι υπάρχει μια μεταστροφή και αυτή η αλλαγή και αυτή η κατάληξη είναι πάρα πολύ σημαντική και πρέπει να τους ευχαριστήσουμε. Επίσης θέλω να ευχαριστήσω την εκπρόσωπο του ΚΟΑΡΜ της, ε, ε, της αρχικής προεδρίας για όλες τις πληροφορίες που μας έδωσε και την ενημέρωση που μας έκανε και χαίρομαι ιδιαίτερα που όλα προχωρούν ικανοποιητικά στην προετοιμασία της συνθήκης ATT. Το θέμα είναι ότι δεν θα πρέπει να είμαστε παθητικοί όσον αφορά την αντιμετώπιση ε, της, των Ηνωμένων Πολιτειών. Ε, αισιοδοξούμε ότι μέσα στα πλαίσια του Γκάτς θα αλλάξει η νοοτροπία και η προσέγγιση των Αμερικανών από την Προεδρία Bush προς την, Προεδρία Ομπάμα. Πιστεύω ότι θα πρέπει να εξασκήσουμε πίεση, να δραστηριοποιηθούμε έντονα ώστε να τους πείσουμε να αλλάξουν στάση. Θα ήθελα να ρωτήσω αν μπορείτε να μας ενημερώσετε για το τι πρόοδο έχουν επιτύχει τα κράτη μέλη ε, στην μεταφορά των διατάξεων της κοινή ε, θέση στην εθνική νομοθεσία. Αν έχετε κάποιο παράδειγμα, αν γνωρίζετε κάτι περισσότερο, διότι υποθέτω ότι όλα τα κράτη-μέλη θα πρέπει τώρα να υιοθετήσουν και να ενσωματώσουν μάλλον την κοινή θέση στην εθνική του νομοθεσία. Ε, και θα πρέπει να προσαρμόσουν τις διαδικασίες τους. Διότι, όπως είπαμε, αυτό το, αυτή η πράξη τώρα είναι νομοθετικά δεσμευτική. Θα ήθελα λοιπόν να ξέρω αν έχετε περισσότερες πληροφορίες. Επίσης, έχουμε εκπρόσωπο της Κομισιόν εδώ. Α, έχουμε, ναι. Ωραία. Θα ήθελα λοιπόν να ξέρω. Τώρα που το Συμβούλιο και η Κομισιόν έχουν δηλώσει την ε, διαφωνία τους επί του θέματος αυτού. Θα ήθελα να ξέρω εάν έχουν την πρόθεση να προσφύγουν στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο. Και θα ήθελα να ρωτήσω το Συμβούλιο και την Κομισιόν τι θα κάνετε, τι, μπορούμε, τι μπορεί να γίνει για να εμποδίσουμε την πώληση ε, ε, ε, όπλων στις χώρες της Αφρικής και την χρήση κονδυλίων του προγράμματος ανάπτυξης του UNDP των, του ΟΗΕ για την αγορά όπλων, παράνομη δηλαδή αγορά όπλων. Είχαμε πολλά παραδείγματα πρόσφατα των τραγικών συνεπειών του, της παράνομης αγοράς όπλων, λαθρεμπορεί όπλων δηλαδή, και οι χώρες ΑΚΕ είναι ομόφωνα εναντίον αυτής της κατάστασης και έχουν τονίσει ότι βασίζονται ιδιαίτερα στην Ευρωπαϊκή Ένωση να υποστηρίξουν την ε, καταπολέμηση αυτού του φαινομένου της, εμπορίας, της παράνομης εμπορίας όπλων. Ο, ο κύριος Ρωμέβα και η κυρία Μπέρ. Θα ήθελα να ολοκληρώσω με τους δύο μιλητές αυτούς τον κατάλογο των ομιλητών, λέει ο πρόεδρος, γιατί έχουμε χρονική, είμαστε υποχρονική πίεση. Ωραία, δύο μιλητές και ολοκληρώνεται, κλείνει ο κατάλογος. Ο κύριος Ρωμέβα. Ε, καταρχήν, ε, ζητώ συγγνώμη που καθυστέρησα. Μπλέχτηκα σε μία διαδήλωση. Ε, πρώτα απ' όλα σας ευχαριστώ που ήρθατε και θα ήθελα να σας κάνω κάποιες ερωτήσεις που κατά γνώμη μου είναι σημαντικές. Πρώτον, ε, θέλω να σας πω ότι με μεγάλη μας χαρά ακούσαμε ότι ο κώδικας συμπεριφοράς εγκρίθηκε ως κοινή θέση και την γνωρίζετε ότι γι' αυτό αγωνιστήκαμε πολύ καιρό. Και η επόμενη ερώτηση είναι συγκεκριμένη. Όσον αφορά τη βελτίωση των κριτηρίων, πού ακριβώ βρισκόμαστε και πώς θα εφαρμόσουμε αυτή την κοινή θέση. Με ποιους όρους και ποιες είναι οι προοπτικές που διανοίγονται μπροστά μας. Ε, πρώτον, σε σχέση με το Ισραήλ και τα συγκεκριμένα βήματα τα οποία πρέπει να γίνουν έτσι ώστε να εμποδίσουμε ε, να φτάσουν όπλα στο Ισραήλ έχοντας κατά νου το ότι διαδραματίζεται τώρα και επίσης και το ότι κατά το παρελθόν ε, δυστυχώς πολλά κράτη ε, παρέδωσαν, εξήγαγαν όπλα στο Ισραήλ. Το τρίτο θέμα που θέλω να ρωτήσω αφορά στις εργασίες για το ATT, τη συμφωνία αυτή Στο θέμα των Ηνωμένων ε, Εθνών ε, υπάρχουν ε, κάποιες εργασίες. Θα θέλαμε να γνωρίζουμε τι είδους προοπτικές έχετε για την εργασία των Ηνωμένων Εθνών επί του θέματος. Και όσον αφορά την τελευταία μου ερώτηση σχετικά με τις εξαγωγές όπλων εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης. Υπάρχει πάντα σχέση ανάμεσα στην εσωτερική και την εξωτερική αγορά όπλων. Και εμείς επανειλημμένα προσπαθήσαμε να το λάβουμε αυτό υπόψη μας. Δεν είμαστε σίγουροι ότι όλα αυτά γίνονται όπως θα το επιθυμούσαμε και ερωτώ κατά πόσον έχετε κάποια νου κάτι πιο συγκεκριμένο όσον αφορά τον έλεγχο της εξαγωγής όπλων. Ähm, Κύριε Μπέα, ευχαριστούμε πολύ για τις πληροφορίες που μας δώσετε. Μία, δύο ερωτήσεις μόνο, δεν έχουμε χρόνο. Πρώτον, όσον αφορά την εξαγωγή όπλων από τη Γερμανία προς το Πακιστάν. Ε, έχω ρωτήσει και την Κομισιόν και το Συμβούλιο πώς αξιολογούν την κατάσταση. Γιατί τότε ε, δεν υπήρχε δεσμευτικός ε, κώδικα συμπεριφοράς και μου απήντησαν ότι τα τελευταία χρόνια δεν έχουν εγκριθεί ούτε ετηθεί εξαγωγές ε, όπλων ε, από γερμανικές επιχειρήσεις προς το Πακιστάν. Βέβαια, λόγω της αλλαγής του δεσμευτικού χαρακτήρα του κώδικα συμπεριφοράς, αν συνέβαινε κάτι τέτοιο θα συνιστούσε παραβίαση εκ μέρους της ε, Γερμανίας. Κατόπιν όσον αφορά την οδηγία περί επιβατών αεροσκαφών. Ε, προφανώς ε, θα γνωρίζετε ενδεχομένως, ρωτώ, έχετε κάνει κάποια ανάλυση κατά πόσο να έχει περιστεί ο έλεγχος ε, παράνομης μεταφοράς όπλων, υπάρχουν αποδεικτικά στοιχεία και αυτά μπορείτε να χρησιμοποιήσετε έτσι ώστε ε, να μπορείτε στο μέλλον να ελέγξετε και καλύτερα την μετακίνηση και το εμπόριο όπλων δια της θαλάσσης. Ε, πολύ ωραία. Κλείνει ο κατάλογος των ομιλητών και το λόγο έχει η ε, κυρία Σεκονισόβα για να απαντήσει. Θα προσπαθήσω να απαντήσω στις ερωτήσεις, τουλάχιστον σε κάποιες εξ αυτών είχαν το ίδιο αντικείμενο. Λοιπόν, ξεκινάω με τον κώδικα συμπεριφοράς που δεν είναι πια κώδικα συμπεριφορά, είναι κοινή θέση. Αλλά ε, κατά κάποιον τρόπο συνεχίζουμε να μιλάμε για κώδικα συμπεριφορά. Πράγματι εγκρίθηκε ως κοινή θέση. Αλλά πρέπει να γνωρίζετε ότι ακόμα και όταν ο κώδικας συμπεριφορά ήταν ένα, μια πολιτική δήλωση δεσμευτική, τα 27 κράτη-μέλη έκριναν τις άδειες εξαγωγής με βάση τον κώδικα συμπεριφοράς. Και όπως γνωρίζετε τα κριτήρια αυτά καθε αυτά δεν άλλαξαν σημαντικά. Σας μίλησα για ε, το κριτήριο υπερθμών 2 που είναι η διεύρυνση έτσι ώστε πλέον να συμπεριλαμβάνεται και το ανθρωπιστικό δίκαιο. Δεν θέλω να σας απογοητεύσω, αλλά παρόλα αυτά πρέπει να σας πω ότι στην καθημερινή εργασία των υπαλλήλων που χορηγούν τις άδειε, δεν θα υπάρξει δραματική αλλαγή με την έννοια ότι επειδή άλλαξε ο κώδικας συμπεριφοράς σε εκείνη θέση θα γίνει κάτι φοβερό. Όχι. Όλοι μας ε, που συμμετέχουμε στις διαδικασίες αδειοδότησης ήδη και κατά το παρελθόν ε, αξιολογούσαμε τις άδειε με βάση τα ισχύοντα κριτήρια. Όσον αφορά τώρα τις εθνικές νομοθεσίες, ε, συζητήσαμε στις άτυπες συναντήσεις στην Πράγα και επίσης και κατά την πρώτη μας επίσημη συνάντηση το Φεβρουάριο. Ορισμένα κράτη-μέλη ήδη εφαρμόζουν τα κριτήρια του πρώην κώδικα και νυν κοινή και τα έχουν συμπεριλάβει αυτά στις εθνικές τους νομοθεσίες. Ορισμένα άλλα κράτη ε, διστάζουν και άλλα πάλι ανακοίνωσαν ότι θα τροποποιήσουν την εθνική τους νομοθεσία. Σύντομα ελπίζουμε έτσι ώστε να εγκριθεί και μία οδηγία για το ενδοκινοτικό εμπόριο, γιατί το θέμα είναι παρεμφερές. Βεβαίως ε, δεν μπορώ να πω σε ποιες χώρες ε, και για πόσο χρονικό διάστημα θα τρέξει αυτή η νομική διαδικασία. Όμως ε, με τη βοήθεια της Γραμματείας του Συμβουλίου ε, θα συγκεντρώσουμε πληροφορίες ε, που θα μοιάζουν με αυτή την κοινή θέση που είχαμε για τη διαμεσολάβηση, για την πρακτόρευση, brokering. Έτσι λοιπόν υπάρχει αυτό το θέμα της ε, υιοθέτησης της ε, νομικής ε, θέσης της εθνικές νομοθεσίες. Τώρα όσον αφορά την κατάσταση στη Γάζα και στη Γεωργία νομίζω είναι κατανοητό ότι οι περιοχές αυτές σας ενδιαφέρουν και προφανώς ενδιαφέρουν όλα τα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Θα γνωρίζετε ότι κάθε συνάντηση της ΚΟΑ ε, γίνεται με τη μορφή γύρου της τραπέζης. Δηλαδή, είμαστε λίγες χώρες, σε λίγες περιοχές και ανταλλάσσουμε εμπειρίες, κυρίως οι χώρες που εξάγουν ε, που κάνουν εξαγωγές σε μια συγκεκριμένη περιοχή. Τα τελευταία χρόνια είχαμε ε, στο γιο τη της τραπέζης και τη Γεωργία και το Ισραήλ. Η Γεωργία το Σεπτέμβριο συγκεκριμένα μετά τα γεγονότα του Αυγούστου Ετέθη ως θέμα λοιπόν η Γεωργία. Η ε, αντιμετώπιση της ε, Γεωργίας ε, τουλάχιστον ε, από τις πληροφορίες που έχω από το Σεπτέμβρη, είναι ότι όλες οι χώρες έχουν παγώσει τις εξαγωγές τους προς τη Γεωργία. Τώρα, για το Ισραήλ είχαμε ε, την τελευταία μας συνάντηση το Φεβρουάριο και ε, από ό,τι φαίνεται συνεχίζονται οι εξαγωγές όπλων προς το Ισραήλ από τα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αυτό έτσι μπορεί κανείς να το δει στην ετήσια έκθεση. Υπάρχουν κάποια άλλα κράτη-μέλη τα οποία όμως είναι αυστηρά, δεν εξάγουν όπλα προς το Ισραήλ και κάποια άλλα το σκέφτονται. Τρεις κατηγορίες κρατών υπάρχουν λοιπόν ε, για τις εξαγωγές όπλων προς το Ισραήλ. Ε, οι εξελίξεις ε, στη Γάζα οδήγησαν ενδεχομένως κάποια κράτη να αναθεωρήσουν τη χορήγηση αδειών. Τώρα, όσον αφορά αυτή τη συμφωνία, την ATT, η εμπλοκή των ΗΠΑ είναι ένα πολύ σημαντικό θέμα όχι μόνο γιατί θέλει κανείς να γνωρίζει την άποψη των κρατών μελών, αλλά και διότι πάρα πολλοί που είναι επιφυλακτικοί και στους οποίους επευθυνθήκαμε κατά τη διάρκεια της εβδομάδας που ήμασταν στη Νέα Υόρκη. Εκεί εξάλλου είχαμε πολλές ε, τρίμερεις ε, συναντήσεις με πολλές ε, αντιπροσωπείες και πολλοί από αυτούς είπαν επανειλημμένα ότι δεν έχει κανένα νόημα εφόσον οι Ηνωμένε Πολιτείε δεν συμμετέχουν. Αυτά όσον αφορά τις άτυπες συναντήσεις της τριμερής. Είχαμε και μία επίσημη ε, τριμερή συνάντηση το Φεβρουάριο. Λίγο μετά την ε, ανάληψη της εξουσίας από τη νέα κυβέρνηση. Και όπως σας είπα και στην αρχή, η θέση των ΗΠΑ για τη Συμφωνία ΕΤΗΤΗ εξακολουθεί να παραμένει ασαφής. Εγώ σας είπα στις εισαγωγικές μου παρατηρήσεις ότι είμαι συγκρατημένα αισιόδοξη. Δεν θέλω να πηδήξω από τη χαρά μου, αλλά εν πάση θέλω να σας πω ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες το σκέπτονται λένε ότι δεν θέλουν να αποδυναμώσουν τους όρους και τα κριτήρια που ήδη ισχύουν με την έγκριση της συμφωνίας γιατί δεν πρέπει να αποδυναμωθούν τα κριτήρια. Αυτό μας απασχολεί και εμάς. Οι συνάδελφοι από τις ΗΠΑ λένε ότι δεν θα θέλαμε να έχουμε μια αιτητή συμφωνία που να έχει αποδυναμώσει τα κριτήρια και παρότι συμφωνούμε για μια συμφωνία αιτητή με συγκεκριμένα κριτήρια. Αυτό δεν σημαίνει βέβαια ότι ορισμένες χώρες δεν μπορούν να έχουν ακόμα πιο αυστηρά κριτήρια για τις εξαγωγές όπλων. Αναγνωρίζουμε λοιπόν τη σημασία της θέσης των ΗΠΑ και βρισκόμαστε κατά κάποιον τρόπο σε συνεχή διάλογο. Αυτό δεν αφορά μόνο την εκάστοτε Προεδρία της Ευρωπαϊκής Ένωσης αλλά και με μονομένα κρατη κράτη-μέλη τα οποία ορισμένα εξ αυτών ε, δραστηριοποιούνται ιδιαίτερα σε τέτοιου είδου θέματα. Νομίζω δεν κατάλαβα καλά την ερώτηση που κάνατε σχετικά με τις εξαγωγές ε, και την εσωτερική και την εξωτερική αγορά. Πολύ θα ήθελα να σε απαντήσω, αλλά δεν ξέρω τι να πω, δεν κατάλαβα καλά. Τώρα, όσον αφορά τα ελαφρά όπλα και τα μικρά, δεν υπάρχει ένα ειδικό κριτήριο που να αφορά στις ε, εξαγωγές ε, στις χώρες ΑΚΕ. γιατί όταν γίνονται εξαγωγές προς αυτές τις χώρες τις ΑΚΕ. Μισό λεπτό, κοιτάξτε, η ερώτηση ήταν τι μπορείτε να κάνετε για να αντιμετωπιστεί αποτελεσματικά το λαθρεμπόριο. Κοιτάξτε, δεν είναι θέμα της ΚΟΑΜ, είναι ένα θέμα καντούν περισσότερο. Αλλά νομίζω ότι και εδώ η συμφωνία ATT παίζει ρόλο. Γιατί αποτελεί ένα σημαντικό κομμάτι των ευρύτερων προσπαθειών αντιμετώπισης του προβλήματος. Επίσης, είπα ότι η απόφαση του Συμβουλίου υπέρ της ATT οδήγησε στο να διοργανωθούν έξι σεμινάρια τον κόσμο. Δύο εξ αυτών στην Αφρική το πρώτο θα λάβει χώρα στο Ντακάρ. για το δυτικό κομμάτι της Αφρικής, αλλά όχι το νότιο και το ανατολικό, για το δυτικό κομμάτι της Αφρικής. Έχουμε λοιπόν ένα πλαίσιο για τα σεμινάρια, αλλά βεβαίως θέλουμε για κάθε σεμινάριο να υπάρχει ένα κεντρικό θέμα και για κάθε περιοχή. Και για τον Ντακάρ σκεφτήκαμε ως ε, κεντρικό θέμα ε, τα ελαφρά και μικρά όπλα. Αυτά είχα να πω. Ευχαριστούμε πολύ, λέει ο Πρόεδρος. Ε, νομίζω ότι τώρα έχει κλείσει ο κατάλογος των ομιλητών. Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω θερμά για την έκθεσή σας. Νομίζω ότι αυτό το το τραγικό, τραγικότατο γεγονός που έλαβε χώρα στη Γερμανία, αυτή η ε, αμόκ κατάσταση που κατέλαβε τον μαθητή δείχνει πόσο σημαντικό είναι να υπάρχουν κανόνες και στο εσωτερικό και στο εξωτερικό σχετικά με τα όπλα. Γιατί το θέμα είναι πρώτον να τηρεί κανείς τους κανόνες και δεύτερον να βελτιώσει ε, τους κανόνες. Νομίζω λοιπόν ότι εδώ ε, κάνουμε ένα σημαντικό βήμα. Το επόμενο είναι εξίσου σημαντικό, ε, δηλαδή αναφέρομαι ε, σε αυτή τη ε, συμφωνία ATT. Και σας εύχομαι καλή επιτυχία στις εργασίες σας και σας ευχαριστώ πολύ που ήρθατε και μας επισκεφθήκατε. Πάμε τώρα στο επόμενο θέμα της ημερήσιας διάταξης, η κυρία Claude France Αρνού, η οποία είναι πρόθυμη να λάβει το λόγο, να μιλήσει. Έχουμε δύο θέματα στην ημερησία διάταξη. Το ένα είναι το chat και τον ε, προπολογισμό του Αθήνα. Έχουμε τσάτ και κεντρικό, κεντροαφρικανική δημοκρατία και τον προπολογισμό του Αθήνα. Ε, θα ήθελα λοιπόν δεν ξέρω αν με καταλαβαίνετε. Καταλαβαίνετε γερμανικά, δεν χρειάζεται ακουστικά. Οπότε φαίνεται με καταλαβαίνετε. Πολύ ωραία. Ε, χαίρομαι λοιπόν που ε, ε, θα έχουμε και την ενημέρωση για τη συνάντηση στο Τσάντ. Ο Γάλλος Υπουργός Εξωτερικών, κύριος Κουσνέρ, μας ε, πρότεινε να χρησιμοποιήσουμε το κυβερνητικό αεροπλάνο της Γαλλίας. Είχαμε λοιπόν τέσσερις ευρωβουλευτές, ε, συνάδελφοι Λαντσμπέργης, ε, Πάσκου, Ινοσκέβιτς ε, και η ταπεινότητά μου. Δύο Γάλλους βουλευτές και ευχαριστώ τον κύριο Ματίσεν γιατί γνωρίζω ότι συνέβαλε στο να διοργανωθεί αυτή ότι η αποστολή του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου που οργανώθηκε και πολύ βραχυπρόθεσμα. Αν μου επιτρέπετε να σας πω εγώ τα δικά μου τα συμπεράσματα από αυτή την επίσκεψη. Ε, αυτή η συνάντηση στο Τσάντ έλαβε χώρα μετά τη Βοσνία Ερσεγοβίνη και ήταν η μεγαλύτερη επιχείρηση που οργάνωσε η Ευρωπαϊκή Ένωση στο πλαίσιο της ε, ΚΕΠΑ. Μέχρι και 3.000 στρατιώτες και στρατιωτίνες. Πάνω από το ίμιση αυτών ήταν Γάλλη, ε, Αυστρία, Ιρλανδία, Πολωνία και εντυπωσιακό αυτό η τρίτη χώρα ήταν η Ρωσία η οποία έστειλε 98 άτομα και 4 ελικόπτερα. Ιδιαίτερα λυπηρό γεγονός κατά την ανάπτυξη αυτής της επιχείρησης ήταν ότι για πρώτη φορά ένας στρατιώτης από ένα κράτος μέλος ε, σκοτώθηκε, ο Ζαν Πολόν κατά τη διάρκεια της επιχείρησης και πρέπει να έχουμε κατά νου ότι προφανώς η Γαλλία τράβηξε, ανέλαβε το μεγαλύτερο ε, βάρος ε, και ο στρατηγός ε, Γκανάσα είχε την ε, ε, γενική την εντολή επιτόπου. Είχαμε και έναν Ιρλανδό διοικητή και αυτό δείχνει ότι ήταν μια διεθνής αποστολή. Ε, εφόσον το πρόσταγμα, το γενικό πρόσταγμα το είχε ένα στρατηγό και υπήρχαν και άλλοι παράλληλα. Είχαμε λοιπόν την ε, δυνατότητα να επισκεφθούμε ένα καταβλισμό προσφύγων και καταβλισμό εκτοπιστέντων. Επισκεφθήκαμε τους πρόσφυγες από τον Νταρφούρ και επισκεφθήκαμε και τον καταβλισμό εκτοπιστέντων από το Τσάντ. Και οι δύο μας είπαν ότι με αυτή την ε, επιχείρηση βελτιώθηκε τα μάλα η δική τους η ασφάλεια, η ατομική ασφάλεια, ε, κυρίως στον καταβλισμό των προσφύγων. Τώρα, όσον αφορά τον καταβλισμό των εκτοπιστένων από το τσάτ αυτό που μας ενδιαφέρει ήταν κατά πόσο οι άνθρωποι αυτοί μπορούν να επιστρέψουν στα χωριά τους. Και εκεί αναφέρθηκαν διάφοροι αριθμοί. Μερικοί είπαν 40.000 ε, επέστρεψαν, άλλοι πάλι είπαν 10.000 επέστρεψαν. Ε, δύσκολο να καταλήξει κανείς κάπου, γιατί υπάρχουν αυτοί που πάνε και έρχονται, που πηγαίνουν έρχονται. Υπάρχουν εκτοπιστέντες που λένε αισθανόμαστε απόλυτα ασφαλείς και τι κάνουν, πάνε πίσω στα χωριά τους, ε, κάνουν τη συγκομιδή και επανέρχονται στον καταβλισμό των εκτοπιστέντων. Γιατί οπωσδήποτε στον, καταβλισμό, στον καταβλισμό με πολύ μεγαλύτερη ασφάλεια από ότι στα χωριά. Όμως ο τελικός στόχος παραμένει οι άνθρωποι να επιστρέψουν στα χωριά του, Βέβαια η ασφάλεια στα χωριά δεν είναι απόλυτη. Εδώ υπολείπονται πάρα πολλά. Αυτό που διαπιστώσαμε ήταν ότι από πλευράς επιμελητίας, επιμελητιακής ε, δομής, ήταν ένα σημαντικό επίτευγμα το να μεταφερθούν όλες αυτές οι δυνάμεις και πρέπει να υπογραμμίσουμε ότι τα στρατεύματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ήταν ευπρόσδεκτα από τους πολίτες, αντιμετωπίστηκαν ως παράγον ασφαλείας. Αυτό λοιπόν το στοιχείο ήταν ιδιαίτερα ε, θετικό. Ε, και πρέπει κανείς επίσης να πει ότι όσον αφορά όλη αυτή τη διαδικασία της αποστολής ε, στρατευμάτων ήταν ε, πολύ χρονοβόρα ε, και το υλικό, τα ελικόπτερα. Εδώ πρέπει να βγάλουμε κάποια συμπεράσματα, να μάθουμε κάποια πράγματα για το μέλλον, γιατί εκεί χρειάζεται κάποια βελτίωση. Ε, παράγον αστάθειας είναι η κατάσταση στο Νταρφούρ. Μέχρι τώρα δεν είδαμε να έρχονται νέοι πρόσφυγες από τον Νταρφούρ. Το γεγονός όμως ότι ο πρόεδρος του Σουδάν εν έχει απαγορεύσει ένα μεγάλο βαθμό λειτουργίας των ΜΚΟ μπορεί να οδηγήσει σε νέο κύμα προσφύγων. Και αυτό ε, μας το εξέφρασαν ως φόβο σε αυτόν τον καταβλισμό. Άρα εδώ υπολείπονται πάρα πολλά για, για τα Έθνη. Εμένα αυτό που με ενδιαφέρε είναι αυτό που είπανε το περίφημο rehatting, αυτό το double hatting, τα δύο καπέλα, τις δύο ε, το έχω ακούσει πολλές φορές, αλλά το re-hatting είναι το εξής οι στρατιώτες από τη Γαλλία, την Ιρλανδία και άλλες χώρες. Έχουμε εκεί στρατιώτες οι οποίοι είναι υπό το πρόσταγμα των Ηνωμένων Εθνών. Και τι κάνουν, αυτοί βγάζουν το καπέλο τους, το βάζουν στην τσέπη και από την άλλη τσέπη βγάζουν άλλο καπέλο και βάζουν και είναι, αντί να είναι στρατιώτες των Ηνωμένων Εθνών, είναι ξέρω εγώ, κάποιου κράτους. Αυτή λοιπόν ε, η αλλαγή του καπέλου ε, μπροστά στα μάτια μας ε, κατέστησε σαφής με απόλυτη, απόλυτα ανάγλυφα. Αυτό που ήταν ενδιαφέρον ήταν ότι θα πρέπει να αναλυφθούν ευθύνες και προς τις δύο κατευθύνσεις. Δηλαδή και όσον αφορά το κοσμοπέδιο, εκεί η Όιλεξ είναι εκείνη που είναι αρμόδια. Στο Τσάντ όμως τα πράγματα λειτουργήσαν αντίθετα. Αυτά αναφέρθηκαν από το διοικητή και είπε επίση ότι σε μελλοντικέ επιχειρήσεις θα μπορούσε κανείς να σκεφτεί πρώτα απ' όλα να στείλει κανείς ε, μία μάχημη δύναμη της Ευρωπαϊκής Ένωσης ε, και κατόπιν να ακολουθήσουν τα Ηνωμένα Έθνη. Για μας ε, αυτό που έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον είναι το θέμα της χρηματοδότησης. Και ο μηχανισμός Αθήνα έχει, είναι ήδη πολύ φορτωμένος ο μηχανισμός αυτός, οπότε θα θέλουμε να αποφύγουμε την περαιτέρω φόρτιση για να μην δημιουργηθούν αδικίες εις βάρος κρατών μελών. Όλα αυτά είναι θέματα τα οποία πρέπει να συζητήσουμε στο μέλλον και γι' αυτό περιμένουμε ανυπομονησία αυτά τα οποία θα μας πει η κυρία Αρνού και σα δίνω αμέσως το λόγο. Mm-hmm. Ε, Πρόεδρε, εσείς ο ίδιος κάνετε τον απολογισμό της ε, όλης επιχείρησης, διότι συμμετείχατε στην ε, παράδοση παραλαβής, παράδοση παραλαβή. Ε, τι να πει κανείς παραπάνω. Ίσως ε, να τονίσω δεδομένου του ότι εγώ συμμετείχα στην διοργάνωση αυτής της επιχείρησης, να τονίζω λοιπόν κάποια στοιχεία. Όπως ε, θα ενθυμίστε, αρχικός στόχος της όλης επιχείρησης ήταν να εφαρμοστούν τα ψηφίσματα των Ηνωμένων Εθνών προκειμένου να αποφύγουμε την περαιτέρω επιδείνωση της κατάστασης μετά από τα όσα συνέβησαν στο Νταρφούρ. Επίσης επιθυμούσαμε να επιτρέψουμε στα Ηνωμένα Έθνη να αναπτυχθούν ειδικά σε ό,τι αφορά σε ζητήματα κατάρτισης των αστυνομικών, χωροφυλάκων κλπ. Και εσείς ο ίδιος λοιπόν πρόεδρε περιγράψατε την βελτίωση στον τομέα της ασφάλειας. Φυσικά δεν μπορεί η βελτίωση, η πρόοδος να είναι θεαματική. Υπάρχουν, υπάρχουν κάποιες χρειές που τονίσατε αναφορικά με τους πρόσφυγες και τους εκτοπιστέντες και τη δυνατότητα επιστροφής τους στα χωριά, αλλά και μη κυβερνητικοί οργανισμοί το αναγνωρίζουν, αλλά και τα Ηνωμένα Έθνη αναγνωρίζουν πως υπάρχει μια βελτίωση στον τομέα της ασφάλειας, κάτι που και εσείς όλοι διαπιστώσατε. Το ότι μπορέσαμε να κάνουμε αυτή τη μεταφορά ε, των εξουσιών, αυτή η παράδοση παραλαβή που έγινε, είναι, αποτέλεσε ιδιαίτερη επιτυχία διότι δεν ήταν διόλου αυτονόητο. Ε, πριν από ένα χρόνο οι αρχές του Τσάντ και οι διάφοροι εταίροι της περιοχής ε, ε δεν έλεπαν με θετικό μάτι την ανάληψη εξουσίας από, την, από τις δυνάμεις του ΟΗΕ αλλά και τις ευρωπαϊκής δυνάμεις που βρίσκεται επιτοπίως. Και αυτό που μας λένε οι συνάδελφοι από τον ΟΗΕ είναι πως υπήρξε ένα θετικό κλίμα λόγω της παράδοσης παραλαβής που έγινε η οποία εξελίχθηκε ικανοποιητικότατα. Και επίσης, όπως είπατε και εσείς, έχει άμεση σχέση με την θετική αντίληψη που είχε ο πληθυσμό. Και εδώ πρέπει να αποτίσουμε φόρο τιμή στους... Δυστυχώς η μιλάει μακριά από το μικρόφωνο. Και ας μην ξεχνάμε ότι χάσαμε και για πρώτη φορά ένα στρατιώτη και χρειάζεται λοιπόν να αποτίσουμε φόρο τιμής και να ευχαριστήσουμε τους ε, στρατιώτες και τη διοίκηση. Ένα στοιχείο που ήταν καθοριστική σημασία και το τονίσατε είναι πως ε, τα περισσότερα κράτη-μέλη τα οποία συμμετείχαν στην ε, επιχείρηση αποφάσισαν να συνεχίσουν τις δραστηριότητε τους υπό την αιγύρια του ΟΗΕ. Αυτό δεν είναι αυτονόητο, υπήρχε δυσκολίε από πλευρά των ε, Ηνωμένων, των Ηνωμένων Εθνών για να συλλέξουν τι διάφορε συνεισφορές των Ευρωπαίων και αυτό το rehiding που είπατε εσείς επέτρεψε να υπάρξει μια μεταβίβαση ε, απόλυτη ηρεμία, κάτι το οποίο επέτρεψε στα Ηνωμένα Έθνη να λειτουργήσουν ικανοποιητικά. Γι' αυτό λοιπόν χρειάζεται να συνεχίσουμε με την... Διότι έχουμε μια, βρισκόμαστε σε μια κατάσταση όπου υπάρχουν κίνδυνοι, υπάρχουν απειλέ και ε, γι' αυτό χρειάζεται και η παρουσία αυτής της πολυεθνική δύναμης. Τώρα να τονίσω το θέμα, κάτι ακόμα το οποίο και εσεί ε, θίξατε Πρόεδρε, είναι το ότι πρόκειται για μια επιχείρηση που ήταν καθαρά ευρωπαϊκού χαρακτήρα, εντάξει υπήρξε μεγαλύτερη εμπλοκή της Γαλλία και αυτό είναι φυσιολογικό διότι τα περισσότερα, περισσότερα μέλη ήταν ε, Γάλλοι. Τώρα τρίτες χώρες ε, και αυτές συνέβαλαν σημαντικά και αυτή είναι η πρώτη ευκαιρία που έχουμε για να υπάρξει συμμετοχή στο ε, διοίκηση και της Ρωσίας. Ήταν λοιπόν μια προσπάθεια σοβαρή, αποτελεσματική. Έχουμε τέσσερα ελικόπτερα ρωσικά και τηρήσαμε τους ε, κανόνες συμμετοχής που συνήθως τηρούμε στην Ευρώπη. Υπήρχαν επίσης και στρατιώτες από την Κροατία και την Αλβανία. Ένα άλλο στοιχείο που είναι πολύ σημαντικό στην όλη επιχείρηση είναι ότι μιλάμε πολύ για μια σφαιρική προσέγγιση. Από την αρχή λοιπόν που έχουμε συμμετάσχει σε παρόμοιες δραστηριότητες φροντίζαμε να μην γίνεται μόνο μια στρατιωτική επιχείρηση αλλά να εντάσσεται πρώτα απ' όλα σε έναν πολιτικό στόχο αλλά και να συνδυάζουμε τα διάφορα μέσα που έχει στη διάθεσή της Ευρωπαϊκή Ένωση και ειδικά το κοινοτικό μέσο. Και αυτή είναι μια προσπάθεια που ήδη από την αρχή μπορέσαμε να συνεργαστούμε με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Η πρώτη fact-finding mission που έγινε στο Τσάντ, οι συνάδελφοι της Κομισιόν προσήλθαν μαζί με το στους εκπροσώπους γραμματείου Συμβουλίου και μπόρεσαν ευθύ εξ αρχής να εντοπίσουν τι μπορεί να γίνει αποτελεσματικά με κοινοτικά μέσα. Κατά τη διάρκεια λοιπόν της όλης επιχείρησης λάβαμε βοήθεια και υποστήριξη από τις μη κυβερνικέ οργανώσεις και εμείς προσθέσαμε να υποβοηθήσουμε το έργο τους στηρίζοντάς τες το τμήμα ανάπτυξης της Κομισιόν επικέντρωσε τις προσπάθειές της δυνατότητα βελτίωσης των συνδικών διαβίωσης στα χωριά από όπου είχαν μετακινηθεί οι πληθυσμοί και με την διεύθυνση ρελέξ της Κομισιόν η οποία σε κονδύλια στην ε, Mirror για τους ε, εκτοπισμένους στο Τσάντ. Υπήρξε λοιπόν μια πολύ καλή συνεργασία στην διαχείριση της κρίσης. Σε κάθε επιχείρηση προσπαθούμε να βελτιώσουμε αυτή τη συνεργασία. Και εδώ πραγματικά νομίζω ότι την πετύχαμε απόλυτα. Νομίζω πως ε, αυτά είναι τα βασικά χαρακτηριστικά της επιχείρησης. Ε, αναφερθήκατε πρόεδρε για τα διδάγματα. Φυσικά θα συνεργάζουμε τα διδάγματα αυτής της επιχείρησης η οποία αποφυλήθηκε φυσικά από τα διδάγματα που είχαμε λάβει από τις προηγούμενες επιχειρήσεις και δει, από το, και δει στο Κονγκό. Θα συνεχίσουμε λοιπόν να εξετάζουμε την κατάσταση και να συνεργάζουμε τα απαραίτητα δάγματα. Εγώ δεν άκουσα την ομιλία του Αλέν Λεωρουά, ο οποίος είχε κάνει τον παραλληλισμό για δύο παραδόσεις ε, που είχαν γίνει στο παρελθόν, παράδοση παραλαβής, αυτό αναφέρομαι. Η συνεργασία μας λοιπόν με τα Ηνωμένα Έθνη είναι πράγματι παραδειγματική διότι πρόκειται για μια συνεργασία που είναι λιγότερο θεσμοθετημένη, αλλά περισσότερο πραγματιστική. Δεν έχουμε κάποιο πλαίσιο, δεν έχουμε κάποιο θεσμικό πλαίσιο. Έχουμε δύο κείμενα ύψη τη πολιτική σημασία, δηλώσει που εγκρίθηκαν υπό Ιταλική και Γερμανική Προεδρία, αλλά είναι μια καθημερινή δουλειά η οποία επικεντρώνεται στι επιχείρησει Η πρώτη στρατιωτική επιχείρηση λοιπόν που αναλάβαμε ήταν η Άρτεμι στο Κονγκό και να στηρίξουμε την Μονίκ την περίοδο όπου η κατάσταση είχε γίνει ανυπόφορη. Λοιπόν, με τα Ηνωμένα Έθνη, είτε πρόκειται στρατιωτικό τομέα, είτε σε πολιτικό, ε, εμείς εστιάζουμε όχι σε θεσμικά ζητήματα συνεργασίας, αλλά σε θέματα ανάγκη συνεργασία. Και η περίπτωση στο Τσάντα ε, ενισχύει την αμοιβαία εμπιστοσύνη και την βεβαιότητα για την συνεργασία υπάρχει μια απόλυτη συμπληρωματικότητα και μπορούμε να εργαστούμε χέρι-χέρι. Κύριε Πρόεδρε, επιτρέψτε να σταματήσω εδώ. Θέλω να σας πω κάτι για το Αθηνά Τώρα ή αργότερα. Αργότερα. Πρόεδρος, ευχαριστούμε πάρα πολύ για την ε, παρουσίασή σας. Εγώ νομίζω ότι αυτή η συνεργασία με τον ΟΗΕ είναι κάτι το οποίο πρέπει να αναπτύξετε. Σίγουρα διαφέρει και τον Αλάν Τιμπουά, ο οποίο είπε ότι η οργάνωση πρέπει να είναι διαφορετική διότι έχουν πάνω από 100.000 στρατιώτες άντρες και γυναίκες σε διαφορετικές επιχειρήσεις. Πάνω από 100.000 και ένα, μια μικρή γραμματεία για την διαχείριση όλων αυτών των στρατιωτών είναι υπερβολικό βάρος πιστεύω χρειάζεται μια μεγαλύτερη ε, γραμματεία και δεν μπορεί και ένας διοικητής να χειριστεί όλα αυτά τα στρατεύματα. Όσον αφορά τώρα τους Ευρωπαίους στρατιώτες, άνδρες και γυναίκες, που ε, δραστηριοποιούνται και για τα Ηνωμένα Έθνη. Αν θυμάμαι καλά είχε πει 1% ήταν οι ε, Ευρωπαίοι στρατιώτες που ήταν και για, τον, για τις εκστρατείες, για τις αποστολές του ΟΗΕ ε, και τώρα έχει ε, σημειωθεί μια αύξηση 200% άρα δηλαδή 3% Ευρωπαίοι στρατιώτες και στρατιωτίνες συμμετέχουν στην, στις δυνάμεις του ΟΗΕ. Είναι υπό τον ΟΗΕ μάλλον ενώ ήταν 1% στο παρελθόν. Ο κύριος Φλίγκερ. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ και για την ενημέρωση που μας κάνετε για αυτή την έκτακτη αποστολή. Εάν θέλουμε να είμαστε ειλικρινείς πρέπει να πούμε ότι ούτε απέτυχε ούτε πέτυχε αυτή η επιστολή. Κάπου ενδιαμέσως κινήθηκε, κάτι ενδιάμεσο ήταν κάτι τάραξε, ταρακουνήθηκαν τα νερά, δεν λέω, αλλά πιστεύω ότι τώρα που ολοκληρώθηκε αυτή η επιστολή θα πρέπει να τα πούμε να μιλήσουμε ειλικρινά και να συζητήσουμε τι γίνεται και γιατί συμβαίνουν αυτά τα οποία γίνονται. Όταν οι 4. παρενέβη οι επιθέσεις κατά ανθρωπιστικών οργανώσεων αυξήθηκαν και η κατάσταση με τους αντάρτες ήταν πάρα πολύ άσκημη. Αργότερα ερέμησαν λίγο τα πνεύματα, αλλά θα ήθελα όσον αφορά αυτή την αποστολή της UFOR υπάρχει το εξής η Γαλλία, εκτός από αυτούς που συμμετέχουν υπό το U4, έχει και δικούς της στρατιώτες. Είναι ένα πολύ πολύ σοβαρό πρόβλημα, διότι αρχικά δεν ήταν, δεν ήταν ξεκάθαρο ποιος ενεργεί, πώς, τι κάνει, ποια δύναμη, η U4 ή η που είναι στη η οι Γάλλοι που είναι της Γαλλίας ας πούμε. Ε, δεν υπήρχε διαφάνεια σε αυτές τις δύο διαφορετικές αποστολές. Αυτό ισχύει ακόμα ε, ε, ε, μέχρι τώρα και το πολιτικό υπόβαθρο ήταν τελείως διαφορετικό Υπάρχει σαφώς αυτό, αυτή η στρατιωτική η συμφωνία, η παραδοσιακή συμφωνία μεταξύ Γαλλίας και Τσάντ. Πάντα υπήρχαν παραδοσιακές σχέσεις και συνεργασίες μεταξύ των δύο αυτών χωρών, ε, Γαλλία και Τσάντ. Και πιστεύω ότι αυτά τα δύο καπέλα των Γάλλων στρατιωτών δημιουργούν προβλήματα και δεν είναι ξεκάθαρη η οριοθέτηση. Ποιες ε, ανθρωπιστικές αποστολές τώρα αποσύρονται, ποιοι είναι αυτοί ε, μάλλον ποιες στρατιωτικές δυνάμεις αποσύρονται, ποιες είναι αυτές που ακόμα υπάρχουν και πόσους στρατιώτες αριθμούν και ποιες ποια ευρωπαϊκά κράτη-μέλη βρίσκονται ακόμα εκεί επί τόπου. Ε, παραθέτω ο, μία έκθεση για το Τσάτ που λέει ότι στο ανατολικό μέρος του Τσάτ θα πρέπει να ληφθούν όλα τα κατάλληλα μέτρα για να αυξηθεί να αναλυφθούν όλα τα μέτρα είναι στο κεφάλαιο 7 για να αυξηθούν οι, οι αποστολές αυτές. Ε, τι εννοούμε τώρα να ληφθούν όλα τα κατάλληλα μέτρα, να ε, ε, στραφούν κατά των ανταρτών, επίσης, απευθείας δηλαδή αντιμετώπιση, αυτό το θεωρώ πολύ προβληματικό πω χτες ε, υπάρχουν υπάρχει κάποια συμφωνία μεταξύ UNAMID και MINOC 2. Έχει γίνει κάποια ρύθμιση συνεργασίας. Επίσης, ε, διάβασα ότι για πρώτη φορά για την αποστολή αυτή χρησιμοποιήθηκε το GMES, δηλαδή το νέο αυτό σύστημα της διορυφορικής επικοινωνίας για να μπορούν να συλλέξουν πληροφορίες. Θα ήθελα λοιπόν να ξέρω αν αυτό το δορυφορικό... Υπάρχουν περισσότερες πληροφορίε για την χρήση αυτού του δορυφορικού συστήματος ε, από πλευράς Κομισιόν. Πιστεύω ότι είναι εξαιρετικά ενδιαφέρον αυτή η δορυφορική πτυχή και θα ήθελα να μάθω περισσότερα. Στο ΩΣΑ και στην Επιτροπή Ανάπτυξης του ΩΣΑ ελέγχθη ότι η στεγιοτική δύναμη στο τσάτ θα πρέπει να θεωρηθεί ως ανα μονάδα δύναμη για την ανάπτυξη της χώρας, για την αναπτυξιακή αποστολή. Άλλο πράγμα στρατιωτική αποστολή, άλλο η αναπτυξιακή αποστολή, άλλο η ανάπτυξη και άλλο για στρατιωτικές ενέργειες. Ποια είναι η θέση της Ευρωπαϊκής Ένωσης έναντι, έναντι αυτής της αναφοράς στην έκθεση του ΟΣΑ της Επιτροπής Ανάπτυξης. Διότι εδώ ε, πρέπει να ε, εφαρμοστούν συγκεκριμένες αναπτυξιακές ενέργειες και θα ήθελα να ξέρω ε, εάν υπάρχει συγκεκριμένος διαχωρισμός μεταξύ στρατιωτικών ενεργειών και αναπτυξιακών δράσεων. Διότι αν μπλεχθούν αυτά τα δύο θα δημιουργηθούν τεράστια προβλήματα. Ας μην ξεχνάμε ότι υπάρχουν και πολλοί αντιφρονούντες οι οποίοι είναι φυλακισμένοι και γι' αυτό ακριβώς δημιουργήθηκε αυτή η, ε, αυτή η έκτακτη κατάσταση κατά την ε, στιγμή που η αποστολή βρισκόταν επί τόπου. Η επίσκεψη γινόταν επί τόπου. Ο κύριος Γκόμες. Η κυρία Γκόμες. Θα, θα ήθελα να σας ευχαριστήσω για αυτή την αποστολή. Τη αποστολή αρχικά είχε κάποια προβλήματα μέχρι να ξεκινήσει. Πρόκειται για μια ευρωπαϊκή αποστολή και υπήρξαν πολλά κράτη τα οποία δεν συμμετείχαν σε αυτήν. αλλά ήταν μια αποστολή δικαιολογημένη, διότι στόχος ήταν να σταθεροποιηθεί μια χώρα που είχε πληγεί ιδιαίτερα από την σύραξη στην γειτονική χώρα, Νταρφούρ και Σουδάν. Άρα. Κατεβλήθη λοιπόν πολύ μεγάλη προσπάθεια από πλευράς επιμελητίας, υπήρξαν πάρα πολλές απαιτήσει και πρόκειται για ένα στίχημα, μια πρόκληση την οποία κερδίσαμε. Επίσης τονίσατε ότι μπορούσε να γίνει παράδοση παραλαβή από το ΟΗΕ μέσα στα προβλεπόμενα χρονικά όρια. Κάτι το οποίο δεν ήταν σίγουρο εξ αρχής. Η παράδοση παραλαβή λοιπόν και όβλουπρας διοίκηση ε, αποτέλεσε ιδιαίτερη επιτυχία. Όλο Όλος ο απόϊχος ο οποίο υπήρξε από ε, μη κυβερνικές οργανώσεις, από πλευράς αρχών του Τσάντ, όλα λοιπόν όσα άκουσα ήταν ιδιαίτερα θετικά σχετικά με την σταθεροποίηση της χώρας αλλά και για θέματα ανθρωπιστικής βοήθειας που χορηγήθηκε στους πρόσφυγες του Νταρφούρ που βρίσκονται στο Τσάντ. Και επίσης θεωρώ πως η όλη επιχείρηση βοήθησε στην σταθεροποίηση του Τσάντ αν και ξέρουμε ότι τα πράγματα παραμένουν ακόμα ιδιαίτερα ρευστά. Και επειδή υπάρχει μια σαφή σχέση ανάμεσα στα όσα συμβαίνουν στο Τσάντ και στο Νταρφούρ και επειδή η σύραξη στο Νταρφούρ συνεχίζει να δημιουργεί σοβαρά προβλήματα λόγω της τάσης των σουδανικών αρχών και της αντίδρασης μετά από την απόφαση του Διεθνούς Ποινικού Δικαστηρίου να καταγγείλει τον πρόεδρο για εγκλήματα πολέμου Ποια είναι η αξιολόγηση των πραγμάτων από πλευρά σας, πώς θεωρείτε ότι μπορεί να εξελιχθούν τα πράγματα και τι γίνεται με τις δυνάμεις που βρίσκονται επί τόπου και κατά πόσον υπεύθυνοι του ΟΗΕ που έχουν αναλάβει τώρα την διοίκηση λαμβάνουν υπόψη όλες τις ε, συνέπειες αυτής της απόφασης του Διεθνούς Ποινικού Δικαστηρίου και των επιπτώσεων που έχει στην περιοχή και στο Τσάντ. Ευχαριστώ. Euh, Να απαντήσω στι ερωτήσει του κ. Φίγκελ. Η κατάσταση αρχικά και η αύξηση στην αρχή και η αύξηση των ε, επιθέσεων. Ρίζα μου πως η κατάσταση ήταν επικίνδυνη και γι' αυτό το λόγο λοιπόν αποφασίσαμε να βρεθούμε. Και τα γεγονότα κατάδειξαν ότι υπήρξαν πάρα πολλές εντάσεις, υπήρξαν επιθέσεις των ανταρτών, το έχουμε λάβει όλα αυτά υπόψη μας κατά τον σχεδιασμό και πραγματικά Αυτή η κατάσταση επηρέασε τις μη κυβερνητικέ οργανώσεις ε, και τις ανθρωπιστικές οργανώσεις. Ε, εντάξει, είπατε ότι δεν πρόκειται για μια καταστροφή ολοκληρωτική, αλλά η κατάσταση έχει βελτιωθεί. Δεν μπορούμε να πούμε, να κάνουμε, να λάβουμε το σενάριο τι θα γινόταν αν δεν είχαμε φτάσει εμείς είναι πιθανότατα η κατάσταση που ήταν ιδιαίτερα ε, ρευστή και επικίνδυνη πριν από την αφήξή μας ε, θα είχε οδηγήσει, θα είχε οδηγήσει σε αποτελέσματα πολύ πιο σοβαρά και καταστροφικά. Τώρα, το θέμα της Γαλλίας. Η Γαλλία έχει παρουσία, είχε μάλλον ανέκαθεν παρουσία στο Τσάντ, όλοι το γνωρίζαμε αυτό, δεν έφτασαν οι Γάλλοι με την αύξηση της Eurofor. μπορούσαν λοιπόν να στηριχτούμε, να βασιστούμε στις ήδη υπάρχουσες γαλλικές δυνάμεις. Η Γαλλία λοιπόν προϋπήρχε στην περιοχή, είχε παρουσία πολλών ετών. Και θεωρώ λοιπόν πως η πολιτική βούληση ε, επιθυμούσε η όλη η δράση να φέρει την ε, ευρωπαϊκή σημαία. Και ο διοικητής ε, των επιχειρήσεων φρόντισε η δράση να είναι ευρωπαϊκή, τηρώντας 100% ε, την εντολή που είχε λάβει η δύναμη, προσπαθώντας ε, να διατηρήσει αμεροληψία, διότι αυτό είναι πάρα πολύ δύσκολο όταν έχετε αντάρτες να σας επιτίθενται και όμως ε, μπόρεσαν να το τηρήσουν. Και επειδή υπήρξε μια συνεχής παρακολούθηση των δραστηριοτήτων του στρατηγού Νάσου, κάτι το οποίο συζητούσε συνεχώς με το ΚΟΠΣ και τους πολιτικούς υπεύθυνους. Ε, φρόντισε λοιπόν όλοι οι παράμετροι της ευρωπαϊκής αυτής επιχείρησης να γίνουν σεβαστές. Και να περάσω κατευθείαν στην ερώτηση που θέσατε για το GMES, που τώρα η Κομισιόν το έχει αναβαπτίσει Κοπέρνικο. Ο Κοπέρνικος λοιπόν δεν ε, ισχύει για τέτοιου είδου ε, αποστολές, είναι μόνο για ε, αποστολές ε, σε μη ναι, στρατιωτικές σε μη, μάλλον σε περιοχές όπου δεν υπάρχει σύραξη και νομίζω ότι αυτή η επιχείρηση στέφεται υπό επιτυχία. Δηλαδή, οι πληροφορίε για πρώτη φορά μπόρεσαν να συνδυαστούν με πληροφορίες που ερχόντουσαν από κυβερνητικό επίπεδο. Ε, από κυβερνητικό επίπεδο. Υπήρξε λοιπόν μια συνεργασία με το Κόσμο Σκανέτ, το Αρλούπε και το Ελίος που θα επιτρέψει στο ε, δορυφορικό κέντρο να λαμβάνει πληροφορίες ε, κυβερνητικής φύσης ε, ε, απόλυτα ασφαλής. Αυτό το οποίο συνέβη στο τσάτ ήταν ακριβώς αυτό το γεγονός και συνδυάστηκε με την συνεργασία όλων των κρατών και το δορυφορικό κέντρο και το κόψο είχε την ευκαιρία να επισκεφθεί τις εγκαταστάσεις στο Μοβαλεριά και στο Τόρεχον και Μπόρεσε λοιπόν στον τομέα της ε, πληροφόρησης ε, μπόρεσε να καταστεί ιδιαίτερα αποτελεσματικό. απέναντι στις της Κομισιόν για το Κοπέρνικο που ε, χρησιμοποιήθηκε ιδιαίτερα για λόγους ανθρωπιστικούς και εγώ χρησιμοποιήσω και το GMS ή το Κοπέρνικο. Πάντως συνεργαζόμαστε να με την Επιτροπή για να δούμε αν υπάρχουν κάποια στοιχεία που μπορούν να συμπεριληφθούν περαιτέρω στον Κοπέρνικο, αλλά το Κοπέρνικος δεν χρησιμοποιήθηκε ως μέσο στήριξη σε μια στρατιωτική επιχείρηση. Είχαμε μέσα κατάλληλα και με μια εντελώς νέα διαδικασία για την χορήγηση πληροφοριών μέσω δορυφόρου για μια επιχείρηση ευρωπαϊκή. Ε, η UNICAT τι πρέπει να κάνει με βάση το κεφάλαιο 7 για τους αντάρτες, δεν καταλαβαίνω καλά τι εννοείται, εάν υπάρξουν επιθέσεις των ανταρτών που θέτουν σε κίνδυνο τους προσφύγους όπου η Unicat θέλει ε, και απαιτείται να τους ε, προστατεύσει, τότε φυσικά μπορεί να χρησιμοποιήσει το άρθρο 7. Οι αντάρτες δεν είναι άνθρωποι που αγωνίζονται <coughs> για κάποιους πολιτικούς λόγους κλπ. Είναι άτομα τα οποία δεν προωθούν τον πολιτικό διάλογο, ούτε τα ανθρώπινα δικαιώματα, ούτε το διάλογο με την αντιπολίτευση. Αυτό λοιπόν που πρέπει να κάνει μια δύναμη, είτε την του είτε της Ευρωπαϊκής Ένωσης, είναι να προστατεύσει τους, τον πληθυσμό Τώρα για το re-hatting, δηλαδή την συνεισφορά των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης στη νέα δύναμη των Ηνωμένων Εθνών. Η πλειοψηφία των δυνάμεων τώρα έχουν τεθεί υπό διοίκηση του ΟΗΕ, δεν ξέρω αν είναι εξαντλητικός ο κατάλογός μου, Αυστρία, Πολωνία, Ιρλανδία, Φιλανδία, Κροατία και Ρωσία. Συμμετέχουν λοιπόν τρίτα κράτη που ήταν μέλη της Eurofor. Συζητήσαμε για να δούμε κατά πόσο θα μπορούσαν και άλλα κράτη να συμμετάσχουν στην αποστολή αυτή. Ε, επέλεξαν να ε, τεθούν υπό τη διοίκηση του ΟΗΕ όπως στην Ορβηγία, κάτι το οποίο θα μπορείς να συνεχίσει στο ρόλο που έπαιζε η Ιταλία στον ιατρικό τομέα. Και ένα τελευταίο στοιχείο, ο συντονισμός ανάμεσα στην Ουνάμι και τη Μινουκάτα λειτουργούσε ήδη στο παρελθόν. Αυτό συνέβαινε ήδη προτού να γίνει η παράδοση παραλαβή. Είναι προφανώς ότι να υπάρχουν δύο δραστηριότητε του ΟΗΕ από τι δύο πλευρέ των συντόρων, αυτό θα διευκολύνει τον ε, συντονισμό. Αυτό που καθιστά την κατάσταση τη Μιναμή δύσκολη και περίπλοκη είναι τα εμπόδια που έχει προκαλέσει η δύναμη αυτή. Και εδώ βλέπουμε τη διαφορά ανάμεσα με την οποία τα ΟΗΕ λειτουργήσε χάρη σε αυτή τη δέσμευση των Ευρωπαίων. Εντάξει, είναι, έχει ιδιαίτερη σημασία αυτό για τον ΟΗΕ, ειδικά για τη συγκεκριμένη επιχείρηση. Δεν μπορώ να σας απαντήσω στην ερώτηση για την Επιτροπή Ανάπτυξης του ΟΣΑ. Αυτό είναι θέμα που αφορά τον ΟΣΑ. Δεν υπάρχει θέση της Ευρωπαϊκής Ένωσης που να προβλέπει ότι οι στρατιωτικές επιχειρήσεις μπορούν να χρηματοδοτηθούν από τον ΟΣΑ διότι δεν ε, είναι επιλέξιμη για βοήθεια, για τη βοήθεια για ανάπτυξη. Εξήγησα προηγούμενα κάποιες ε, δράσεις που αφορούν συγκεκριμένα την τομέα της ανάπτυξης και στο Τσάντ. Αυτό το προσπαθήσαμε. Και τα κράτη-μέλη προσπάθησαν να αναπτύξουν όπως το έπρεξε και η Κομισιόν μια αναπτυξιακή δράση γύρω από τις δραστηριότητες ε, των επιχειρήσεών της. Ε, σε ό,τι φορά τα πολιτικά προβλήματα απάντησα. Αυτό ήταν σταθερό μέλημα της Ευρωπαϊκής Δράσης και αυτό που έγινε στο ειδικό επίπεδο προχώραγε χέρι-χέρι με μια πολιτική δραστηριότητα προκειμένου να ευνοήσουμε τον διάλογο με την αντιπολίτευση, να παροτρύνουμε την κυβέρνηση του Τσάντα προς ε, μια στάση και μια συμπεριφορά που ανταποκρίνεται στα πρότυπα τα ευρωπαϊκά και αυτή είναι μια δράση η οποία θα συνεχιστεί. Όπως επίσης η δράση που αναλάβουμε σε ανθρωπιστικό επίπεδο και σε επίπεδο αναπτυξιακό δεν ε, έχουμε φτάσει στο τέλος της ε, δραστηριότητάς μας στην περιοχή των Αντίων. Τώρα παντώντας την κυρία Γκόμες, ποια είναι η αξιολόγηση των επιπτώσεων της κατάστασης στο Σουδάν. Φυσικά αυτό ήταν ένα μέλημά μας εδώ και χρόνια. Συζητούσαμε με τον ΟΗΕ για τον κίνδυνο ο οποίος μπορεί να προκύψει από την κατηγορία του Προέδρου ως εγκληματία πολέμου. Τώρα υπάρχει αυτή η απαγόρευση προς ανθρωπιστικές οργανώσεις να κάνουν τη δουλειά τους παρακολουθούμε τις εξελίξεις ε, με μεγάλη προσοχή. Δεν υπάρχουν προς το παρόν άμεσες επιπτώσεις στο Τσάντ ε, και ειδικά για τους πρόσφυγες είναι προφανές ότι τα Ηνωμένα Έθνη έλαβαν αυτό υπόψη τους στον όλο και εμείς επίσης το λάβαμε υπόψη στον σχεδιασμό της ε, μεταβατικής περίοδου. Ευχαριστώ. Θα ήθελα και εγώ να προσθέσω δύο να κάνω δύο παρατηρήσεις. Καταρχάς για την ε, αντικειμενικότητα της u του U4 ε, και πρέπει αυτό να ληφθεί πολύ σοβαρά υπόψη γιατί ήταν και ένα από τα αιτήματα της Γαλλίας. Καταρχάς, ε, ένα από τα στοιχεία τα οποία έχουν επιφέρει σοβαρές επιπτώσεις είναι ότι υπάρχει πετρέλαιο στην περιοχή και το πετρέλαιο αυτό βεβαίως δεν το εκμεταλλεύεται καμία γαλλική εταιρεία αλλά μία αμερικάνικη και πολλές κινέζικες εταιρείες. Αυτό είναι ένα επιπρόσθετο επιχείρημα. Δεύτερον, ο Κοπέρνικος και το θέμα του δορυφορικού κέντρου. Είχαμε πάντοτε πιέσει έντονα ότι είναι αναγκαίο οι εικόνες ε, των τρίων αυτών οργανώσεων ε, της, της, της γερμανικής, γαλλικής ε, και της τρίτης πλευράς να είναι στη διάθεσή μας μέσω δορυφόρου. Οι εικόνες αυτές λοιπόν να είναι διαθέσιμες μέσω δορυφόρου. Αυτό πράγματι συμβαίνει ε, και είναι διαθέσιμες στις τρεις ε, συμμετέχουσες πλευρές. Όταν λοιπόν στέλνουμε στρατιώτες ή στρατιωτίνες είναι πολύ σημαντικό να έχουμε και αυτήν την ενημέρωση, ε, τη δορυφορική ενημέρωση για να μπορούμε να καλύψουμε τις ανάγκες. Είπαμε λοιπόν στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ότι... Α, συγγνώμη, μπερδεύομαι εδώ. Ο, Κο... Ο Κοπέρνικος κατά την άποψή μας ανήκει, ανήκει μέσα σε αυτές τις προδιαγραφές. Υπάρχει κανείς από την Κομισιό να μας εξηγήσει πώς ακριβώς έγινε αυτή η ρύθμιση. Όχι. Δεν υπάρχει. Όμως αυτό είναι ένα ερώτημα που μας ενδιαφέρει. Στο πλαίσιο του Γαλιλαίου είχαμε επιτύχει μια ευρεία συνένεση και είχαμε πει και το σύστημα του Γκαλιλαίου θα πρέπει να είναι διαθέσιμο για στρατιωτικές και μη επιχειρήσεις όπως συμμετέχουν ευρωπαϊκές δυνάμεις. Δηλαδή το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο με μεγάλη υπερψηφία είχε εκφράσει την άποψή του ότι αυτά τα τεχνικά μέσα που διατίθενται θα πρέπει να ε, διατίθενται ε, και μέσα στο πλαίσιο της ΚΕΠΑ. Ο κύριος Γιανοβιέτσκι. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ζητώ συγγνώμη, κυρία Διευθύντρια, διότι θα ήθελα να θέσω και εγώ μια ερώτηση που ήδη ετέθη, που είναι ένα ζήτημα αρκετά σημαντικό για την περιοχή. Εντάξει, δεν είναι δική σας ευθύνη, αλλά είναι κάτι που μας συγκλονίζει. Δηλαδή το πρόβλημα του του, Σουδάν. Τι πιστεύετε. Εμείς θέλουμε να επιλύσουμε το πρόβλημα, θέλουμε να αποσταρρεύσουμε τον πληθυσμό, να βοηθήσουμε τους πρόσφυγες. Εγώ δεν είμαι κατά του ποινικού δικαστηρίου και κατανοώ πως πρέπει να εφαρμοστούν αυστηρά μέτρα για τους ανθρώπους που παραβιάζουν τον νόμο ή διώκουν πληθυσμούς. Το πρόβλημα όμως μπορείτε να το κοιτάξετε εκ του σύναγκης. Γνωρίζετε πολύ καλύτερα το πρόβλημα από ότι εμείς. Θεωρείτε λογική λοιπόν αυτήν την ε, δίωξη του Προέδρου με τις ε, δυνατότητες τώρα που έχουμε παρέμβαση ε, στο Σουδάν. Κύριε Αρνού. Ναι, πολύ καλά καταλάβατε ότι με ξεπερνάει αυτό το θέμα, δεν είναι στις δικές μου ευθύνες. Μπορώ να σας μιλήσω, μάλλον προτιμώ να σας μιλήσω για θέματα που γνωρίζω. Όλοι θεωρώ ότι γνώριζαν την κατάσταση. Υπάρχει διεθνής δικαιοσύνη, διεθνές δίκαιο που θέλουμε να εφαρμοστεί, αλλά ξέρουμε ότι μπορεί να έχει και κάποιες επιπτώσεις, όπως έχετε και εσείς κατά νου. Όλοι νομίζω το έχουν κατά νου αυτό. και σίγουρα το σκέφτηκαν πριν πάρουν την απόφαση, αλλά δεν μπορώ να σα απαντήσω να σα πω περισσότερο. Πρόεδρε, μου επιτρέπετε, μια που δεν απάντησε η Κομισιόν για τον Κοπέρνικο, γιατί αναφερθήκατε στο ενδιαφέρον που έχει το Κοινοβούλιο στο να γίνει καλή χρήση των μέσων που διαθέτουμε σε ε, επίπεδο διαστημικό. Ε, Υπάρχει λοιπόν στενή συνεργασία μεταξύ, συμβουλίου, ε, μεταξύ Κομισιών και Κοινοβουλίου για τα θέματα του διαστήματος και το ε, διαστημικό κέντρο ήδη συνεργάζεται για ορισμένες πτυχές αυτό το τορεχόν το κέντρο ε, συνεργάζεται με την Κομισιόν σε θέματα που αφορούν το GMS Κοπέρνικο και με την ε, Κομισιόν εξετάζουμε πώς ε, αυτά τα, αυτό το κέντρο θα μπορούσε να υποστηρίξει περαιτέρω τον Κοπέρνικο. Και εμεί για την επιχείρηση χρησιμοποίησαμε εικόνες που βρίσκονται από ένα σύστημα διαφορετικό από το Έλιους και το Διαστημικού Κέντρο. Θα ήθελα να πω ότι ε, όλα αυτά τα στηρίζει η πλειοψηφία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Κοιτάξτε, εγώ ε, προσωπικά είδα τα υπέρ και τα κατά και πρέπει να σας πω ότι συνηθίζω να μιλάω μόνο για πράγματα που δεν έχουν ακόμα αποφασιστεί. Αυτό το θέμα όμως κρίθηκε ήδη. Δηλαδή το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο έλαβε την απόφασή του και τώρα εκείνο που τίθεται το θέμα είναι ε, πώς ε, τι τοποθετούμεθα εμείς σε αυτήν την απόφαση και πώς ε, θα κατορθώσουμε στους ε, καταβλισμούς ε, προσφύγων να δημιουργηθούν οι σωστές συνθήκες διαβίωσης και από την άλλη να συνεχίσουμε να καταβάλουμε προσπάθειες έτσι ώστε η διένεξη αυτή να επιληθεί σε πολιτικό επίπεδο γιατί στρατιωτικά δεν μπορεί να κρυθεί αυτή η σύγκρουση δεν υπάρχει καμία τέτοια πιθανότητα η κυρία Γκόμες Πρόεδρε, μία διευκρίνηση. Δεν θα ήθελα η ερώτηση που έθεσα για το θέμα της, ε, των κατηγοριών απέναντι στον πρόεδρο Μπασίρ να προκαλέσει κάποιες εμβολίες σχετικά με το ε, Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο. Αναμφίβολα το δικαστήριο έχει τους λόγους του είναι βάσιμη για να προβεί σε κάτι τέτοιο. Και Εμείς πρέπει να βοηθήσουμε προκειμένου να συλληφθεί και να οδηγηθεί στην δικαιοσύνη αυτό το άτομο. Η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει εργαστεί ώστε το ζήτημα του Νταρφούρου να, να μεταφερθεί στο ποινικό διεθνές δικαστήριο, διότι το Σουτάντα δεν αναγνώρισε ποτέ την ε, δικαιοδοσία του Διεθνούς Ποινικού Δικαστηρίου χάρη στην εργασία, στη συνεργασία μάλλον της Ευρωπαϊκής Ένωσης και αυτό το ξέραμε πολύ καλά με την, όταν υπήρχε η κυβέρνηση Μπούς στις ΗΠΑ που μέχρι τώρα δεν αναγνώρισε την δικαιοδοσία του Ευρωπαϊκού Διεθνούς, του Διεθνούς Ποινικού Δικαστηρίου. Λοιπόν, εάν ενεργεί τώρα το δικαστήριο. Αυτό είναι αποτέλεσμα της προσπάθειας που έχει καταβάλει η Ευρωπαϊκή Ένωση. Δεν υπάρχει περίπτωση λοιπόν η Ευρωπαϊκή Ένωση να θέσει ένα αμφιβόλο την απόφαση αυτή του Διεθνούς Ποινικού Δικαστηρίου. Πρόεδρος, ε, ο κύριος Φλούδια, για ένα μόνο λεπτό το γεγονός ότι σχολιάσατε κι εσείς, αυτό δημοκρατικά σωστό είναι. Αυτό ήθελα να το πω. Αυτό που έχει ενδιαφέρον για μένα είναι ότι δεν λέει τίποτα η Κομισιόν. Νομίζω ότι αυτό δεν μπορούμε να το καταπιούμε ως Κοινοβούλιο, γιατί εδώ πρόκειται για ένα σημαντικό θέμα. Είναι ξεκάθαρο. Κατά τα άλλα, η νομική βάση είναι σαφής. Λέει, και το είπε για άλλη μια φορά η ομιλήτρια, η νομική βάση αναφέρει και εδώ το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο μπορεί να αποφασίσει ότι θέλει. Μόνο που η νομική βάση λέει ότι η χρήση μπορεί να είναι καθαρά και μόνο πολιτική. Ε, εφόσον λοιπόν ε, δεν υπάρχει ακόμα η συνθήκη της Λισαβόνας, δεν ανάγκη να γίνεται αυτή η συζήτηση. Υπάρχει μια νομική βάση και πρέπει να τοποθετηθούμε πάνω σε αυτήν. Ε, Γι' αυτό ε, λοιπόν ε, η στάση σχετικά με τις ε, στρατιωτικές αποστολές είναι προβληματική. Εγώ θα ήθελα να ακούσω κάτι από την Κομισιόν όπου βέβαια το θέμα δεν είναι δικό μας ούτε του Συμβουλίου ούτε δικό μας είναι της Κομισιόν. Πρόεδρος, λαμβάνω υπόψη μου αυτά που είπατε για τη νομική βάση και εν ευθέτω χρόνο θα πρέπει να εμβαθύνουμε. Θα έλεγα Τώρα ε, να περάσουμε στο θέμα Α, Αθήνα. Πολύ ωραίο το όνομα. Πάμε τώρα στη Θεά Αθήνα και επ' αυτού θα ήθελα να δώσω το λόγο στην κυρία Αρνού. Ευχαριστώ πρόεδρε. Η Αθηνά συστάθηκε προκειμένου να διευκολύνουμε την διαχείριση μια επιχείρηση όπω γνωρίζετε, οι συνθήκε τη Ευρωπαϊκή Ένωση προβλέπουν σε ό,τι φορά τι επιχειρήσει που έχουν επιπτώσει επιπτώσεις ε, αφορούν στο τομέα τη άμυνα, η χρηματοδότηση είναι χρηματοδότηση μέσω κρατικών συνεισφορών, όχι δηλαδή μέσω του κοινωνικού προπολογισμού. άρθρο 28.2 του συνθήκης, νομίζω το γνωρίζετε. Τώρα, για να διευκολύνουμε την εφαρμογή αυτών των στρατηγικών δραστηριοτήτων της αρχής του 2004 ε, εφαρμόσαμε το μηχανισμό Αθηνά για τη διαχείριση του κοινού κόστους των επιχειρήσεων αλλά η χρηματοδότηση αυτή παραμένει χρηματοδότηση που έρχεται από τη συνεισφορά των κρατών μελών και που υπολογίζονται με βάση το εθνικό ΑΕΠ Επιτρέπει λοιπόν να αναλαμβάνουμε το κοινό κόστος που αφορά το στρατηγείο και τις υποδομές και δεύτερον τη χρηματοδότηση των ε, κοινών δράσεων ανάλογα με την κατανάλωση των κονδυλίων. Λοιπόν, στην αρχή τη ε, επιχείρηση υπολογίζουμε ένα ποσό που είναι μια εκτίμηση του κοινού κόστους για μια συγκεκριμένη επιχείρηση και έπειτα το Συμβούλιο εγκρίνει τον προϋπολογισμό της όλης επιχείρησης με βάση τις, τα έξοδα των πρώτων μηνών. Αυτή λοιπόν η αρχή του Αθηνά ως πλεονέκτημα επιχειρησιακά επιτρέπει να γίνει η σωστή κατανομή των δαπανών, επιτρέπει καλύτερη λειτουργία τους της όλης προσπάθειας, της όλης επιχείρησης και επίσης μέσω ενός συστήματος που ενός ζητήματος χρηματοδότης. Και αυτό είναι ένα στοιχείο κλειδί, δηλαδή πρέπει ευθύ εξ αρχή να έχουμε ένα σύστημα το οποίο θα μας επιτρέπει να συλλέγουμε, να συγκεντρώνουμε μάλλον τα απαραίτητα ποσό, τα ποσά για τις υποδομές και για, το, για όλο το υλικό. Αυτό λοιπόν είναι το σύστημα Αθηνά, είναι ένα σύστημα ευέλικτο ρεαλιστικό θα έλεγα διότι λαμβάνει υπόψη το γεγονός ότι η συνθήκη προβλέπει πως σε αυτό τον τομέα έχουν στρατιωτικές δραστηριότητε και αμυντικές δραστηριότητε και παραμένει η χρηματοδότηση και η χρηματοδότηση μάλλον γίνεται από τα κράτη-μέλη αυτό λοιπόν ήταν το πνεύμα της συνθήκης και αυτή η συνθήκη θα πρέπει να γίνει σεβαστή. Γι' αυτό λοιπόν προβλέπεται αυτό η χρηματοδότηση Αθήνα διεξάγονται συχνά έντονες συζητήσεις αναφορικά με το τι είναι κοινό κόστος και τι όχι. Ε, π.χ. παρατείναμε το σύστημα που μας επιτρέπει να διατηρήσουμε για τις ομάδες μάχης, τις μάχημες ομάδες ε, ένα κόστος ε, ευρύτερο, μεγαλύτερο π.χ. για τη δυνατότητα μεταφοράς ε, με αεροπορικής ε, κάποιων στρατευμάτων, άμα είναι μονάδες ε, για μια γρήγορη ανάπτυξη, ταχύες ανάπτυξης. Αυτές οι ρυθμίσεις ισχύουν μέχρι τα τέλη 2009. Σας ανέφερα μερικές αρχές, γενικές αρχές του Αθηνά. Εάν έχετε ερωτήσεις, ο συνάδελφός μου Τιέρι Μπουσέ και εγώ είμαστε στη διάθεσή σας. Ε, θα ήθελα να ρωτήσω κάτι. Δηλαδή, σε κάθε επιχείρηση υπάρχουν χώρες οι οποίες ε, απέχουν και μετά υπάρχουν χώρες οι οποίες ε, συνενούν. Λένε όμως ότι δεν θα συμμετάσχουν και υπάρχουν και άλλες χώρες οι οποίες συμμετέχουν. αυτή είναι η κατάσταση. Τώρα, εγώ ερωτώ, αυτός ο μηχανισμός, ε, ο μηχανισμός ε, Αθηνά αφορά και εκείνες τις χώρες που έχουν δηλώσει αποχή, αφορά και εκείνες τις χώρες που λένε ναι θα συμπράξουμε, μάλλον συμφωνούμε, αλλά δεν θέλουν να συμμετάσχουν ή αφορά μόνο τις χώρες εκείνες που συμμετέχουν σε μια επιχείρηση. Ο μηχανισμός Αθηνά εφαρμόζεται σε όλα τα κράτη-μέλη πλην της Δανίας που έχει δηλώσει opt-out. Ό,τι είναι κοινό λοιπόν αναλαμβάνεται από κοινού. Υπάρχει μια θεωρητική διάταξη που επιτρέπει σε μια χώρα μέλος να απέχει και άρα να μην συμμετέχει στην κοινή χρηματοδότηση. Αλλά αυτή η διάταξη δεν έχει ποτέ χρησιμοποιηθεί μέχρι τώρα. Υπάρχει όμως τη συνθήκη. Υπήρξαν ε, αρκετοί που εξεπλάγησαν από το γεγονός ότι παρόλα αυτά ε, χώρες ε, που συμμετείχαν στη χρηματοδότηση δεν θέλησαν να συμμετάσχουν στην πραγματική επιχείρηση. Ίσως βέβαια να μην είδαν το κείμενο, λέει ο Πρόεδρος. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, με πάση περιπτώσει, για τη διευκρίνηση. Άρα δηλαδή θεωρητικά υπάρχει δυνατότητα μια χώρα να δηλώσει αποχή και όταν το κάνει αυτό δεν χρειάζεται να πληρώσει. Έτσι δεν είναι. Πολύ ωραία. Σας ευχαριστώ πολύ. Ο κύριος Φλούγκα. Κοιτάξτε, εγώ νομίζω ότι τώρα μόλις ε, θίξατε ένα ιδιαίτερα σημαντικό θέμα. Γιατί ας πούμε στην συγκεκριμένη περίπτωση Τσάτ και Γερμανία. Η Γερμανία πλήρωσε από ό,τι ξέρω και ε, την ε, πληροφορία που δώσατε τη βρήκα πολύ ενδιαφέρουσα όμως δεν αντιστοιχεί με αυτά που ξέρω εγώ μέχρι τώρα, τουλάχιστον εμπειρικά. Αν ισχύει αυτό που λέτε εσείς, καλώς. Εγώ είχα καταλάβει ότι η Δανία, λόγω ακριβώ της ρήτρας αυτοεξαίρεσης, μπορεί να μην συμμετάσχει στη χρηματοδότηση. Ε, το θέμα είναι πράγματι θα ήταν πολύ ενδιαφέρον να δούμε τι ακριβώ γίνεται με αυτές τις τρεις κατηγορίες που έθιξε ο κύριος Φων Βόγκαου η βιβλιογραφία επί του θέματος είναι ιδιαίτερα αντιφατική και χρειαζόμαστε μια ξεκάθαρη άποψη. Υπάρχει κάποια δυνατότητα για ένα κράτος μέλος να πει δεν πληρώνω. Η κοινή δράση το προβλέπει. Υπάρχει περίπτωση της Δανίας που εξορισμού έχει επιλέξει το opt-out και δεν συμμετέχει. Αυτό είναι αυτόματο. Κατά ε, τα υπόλοιπα, ο κανόνας είναι πως όλα τα κρατημέλη συμμετέχουν στο κοινό κόστος είτε συμμετέχουν είτε όχι στην επιχείρηση. Κάτι το οποίο δεν είναι τόσο υψηλό, δεν υπάρχει ιδιαίτερη αλληλεγγύη θα έλεγα. Το κοινό κόστος είναι ένα μικρό κομμάτι της δαπάνης. Κατά ε, τα υπόλοιπα είναι όπως το ΝΑΤΟ. Ισχύουν τα αυτά. Δηλαδή όσοι, όσοι συμμετέχουν πληρώνουν. Αυτό είναι ένα μικρό κομμάτι της όλης αλληλεγγύης που εκφράζουν τα κράτη-μέλη όταν έχει αποφασιστεί η ανάληψη δράσης. Και η άλλη περίπτωση είναι όπου ένα κράτος μέλος αναγγέλει εκ των προτέρων πως θα απέχει και άρα δεν θα συμμετάσχει και στην κοινή χρηματοδότηση. Είναι μια δυνατότητα που προβλέπεται στην συνθήκη γενικά και άρα μπορεί να εφαρμοστεί και στην Αθηνά. Σας ευχαριστώ πολύ. Η κυρία Γκόμες. Όπως είπε η κυρία Αρνού, νομίζω ότι το κομμάτι που καλύπτεται από το κοινό κόστος ε, αντιπροσωπεύει περίπου το 10% της ε, συνολικής δαπάνη ε, μιας επιχείρησης. Νομίζω ότι αυτό είναι ένα σημαντικό μειονέκτημα. Θα πρέπει να δούμε λοιπόν πώς θα μπορούσαμε να διευρύνουμε το, ορισμό του κοινού κόστους έτσι ώστε να υπάρξει μεγαλύτερη συμμετοχή στην χρηματοδότηση. Και η χρηματοδότηση των αποστολών αυτών να μην καθυστερούν ή να παρεμποδίζουν την ε, ανάπτυξη της ε, επιχείρησης, της αποστολής. Τι πιστεύετε ότι εμείς μπορούμε εδώ στο Κοινοβούλιο να κάνουμε ώστε να βοηθήσουμε για να συμφωνήσουν τα κράτη-μέλη σε έναν ορισμό ευρύτερο για το τι εντάσσεται μέσα στο κοινό κόστος. Όπως γνωρίζετε αυτό είναι ένα ζήτημα περίπλοκο οι θέσεις των κρατών μελών είναι πολύ διαφορετικές. Ως Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο φυσικά έχετε κάθε ελευθερία και μπορείτε να εκφράσετε την επιθυμία μεγαλύτερη αλληλεγγύη και αποτελεσματικότητα. Επίσης και σε εθνικό επίπεδο είναι σημαντικό να διεξαχθεί η πολιτική συζήτηση ε, φυσικά δεν εμπίπτουν στις δικές μου αρμοδιότητες, μια πολιτική συζήτηση για να δούμε κατά πόσο στις πρωτεύουσες ε, επιθυμούν να υπάρξει μια αλληλεγγύη όταν, όταν γίνονται τέτοιες ε, δραστηριότητες φυσικά πρέπει να συζητηθεί θέμα και στο επίπεδο του ΝΑΤΟ ήδη διεξάγεται μια συζήτηση εκεί και υπάρχει μια τάση προκειμένου να υπάρξει μεγαλύτερη συμμετοχή του κοινού κόστους δεν θα ήταν καλό για την Ευρωπαϊκή Ένωση να συμβεί κάτι τέτοιο χωρίς αυτή να υποφεληθεί από μια ανάλογη αύξηση διότι το κράτος μέλος που θα στείλει μια μάχημη μονάδα θα αναλάβει ένα υψηλότερο κόστος όπως είπατε και εσείς οι αποφάσεις συλλαμβάνονται με ομοφωνία και το κοινό κόστος είναι ένα μικρό κομμάτι της όλης επιχείρησης. Σας ευχαριστώ πολύ. Ήταν μια σημαντική συζήτηση για μας, αυτή την οποία κάναμε και ε, απαντήθηκαν πολλά ερωτήματά μας. Θα πρέπει λοιπόν να εξετάσουμε δύο θέματα. Πρώτον, την μη στατιωτική συνεργασία και την κατανομή των βαρών για την μη στρατιωτική συνεργασία και δεύτερο την ρύθμιση των λεπτομεριών, δηλαδή την εμβάθυνση του, του προγράμματος Αθήνα και τι ανήκει, τι καλύπτεται από το πλαίσιο Αθήνα και δεν καλύπτεται. Ε, οι λεπτομέρειες είναι πολύ τεχνικές, όμως δεν μπορούμε να αποφύγουμε ε, την εμβάθυνση σε αυτό το ζήτημα και πιστεύω ότι ε, είναι και πολύ ενδιαφέρον να δούμε ακριβώς τις λεπτομερείς πτυχές της χρηματοδότησης και της συγχρηματοδότησης. Αν δεν υπάρχουν άλλοι ομιλητές επί του θέματος, τότε θα ήθελα να ευχαριστήσω θερμά την κυρία Αρνού για αυτή τη συζήτηση και την επιτυχή συνεργασία μας. Και είστε, έτσι εύχομαι, στο Ιπανιδίν. Και προχωρούμε τώρα στην ε, συζήτηση για τη γεωργία. Τα ανταλλαγή απόψε. Σημείο 7. Ε, μπορούμε, πιστεύω, να είμαστε σύντομοι σε αυτό το θέμα. Όμως, ε, πρέπει να ενημερωθούμε μετά από την επίσκεψη που κάναμε στη Γεωργία και τα ε, γεγονότα τα οποία διαπιστώσαμε και πιστεύω ότι με τις σημερινέ συνθήκες η Ευρωπαϊκή Ένωση έκανε μια πολύ επιτυχημένη ε, και, και οργάνωσε μια επιτυχημένη αποστολή και μάλιστα ταχύτατα και θα ήθελα να ευχαριστήσω και τη Γραμματεία του Συμβουλίου για τη συνεργασία. Πιστεύω ότι ήταν μια κατεπίγουσα ε, ενέργεια αυτή ε, και αυτή η μη στρατιωτική ε, δράση έδειξε ότι μπορούμε να αναλάβουμε και να διοργανώσουμε κάτι γρήγορα όταν υπάρχει ανάγκη. Αυτό δεν σημαίνει ότι δεν ε, ξεκολουθούν να υπάρχουν πάρα πολλές ε, δυσκολίες. Οι παρατηρητές μας ε, δεν μπόρεσαν να προχωρήσουν περαιτέρω προς την Απχαζία και άλλες περιοχές. Από τη μία πλευρά έχουμε προ, προωθημένες, πρέπει να πείσουμε προωθημένες θέσεις ε, διαφόρων μονάδων και από την άλλη πλευρά οδοφράγματα ε, τα οποία μας εμποδίζουν να προχωρήσουμε, να μπούμε στην επικράτεια, στα, στα εδάφια αυτά όπου έχουν γίνει μεγάλες καταστροφές ή δεν, δεν μπορέσαμε τουλάχιστον η διεισόμαση να διαποστώσουμε εμείς τις τεράστιες αυτές καταστροφές όπως λέχθη αυτό το οποίο όμως διαπιστώσαμε είναι ότι οι πολιτοφύλακες δηλαδή οι πολίτες που ήταν ντυμένοι με στατιωτικά ρούχα θα πρέπει και αυτές, ε, και αυτές οι δυνάμεις των, της πολιτοφυλακής να ληφθούν υπόψη. Ε, ε, και ο κύριος ο συνάδελφος Χάουτ ήταν εκεί και συζητήσαμε και το τι βοήθεια μπορεί να προσφερθεί μέσα στα πλαίσια του ΩΣΑ. Ε, είπαμε ότι μόνο η Ευρωπαϊκή Ένωση θα είναι ε, πλέον εκεί, θα εκπροσωπείται εκεί, οπότε τίθεται και το θέμα της ε, χρονικής προθεσμίας, για πόσο χρονικό διάστημα δηλαδή θα παραμείνει εκεί αυτή η δύναμη όταν πλέον δεν θα δραστηριοποιούνται άλλες, άλλοι οργανισμοί, φορείς όπως ο ΩΣΑ Και ότι εάν είχαμε, είχαμε τη δυνατότητα να επισκεφθούμε τις δύο αυτές επαρχίες, έστω και από περιορισμένες συνθήκες, θα είχαμε διαπιστώσει περισσότερα πράγματα, δεν μπορέσαμε όμως να το κάνουμε και γι' αυτό θα μας απασχολήσουν αυτά τα συγκεκριμένα εδάφη και στην επόμενη θητεία του σώματος. Θέλει κανείς να μιλήσει επί του θέματος. Mr. Θα ήθελα καταρχάς να σας ευχαριστήσω, Πρόεδρε, για την ε, εξαιρετική διοργάνωση αυτής της αποστολής. Πιστεύω ότι ήμασταν λίγαν αποτελεσματικοί, εκτελέσαμε πολύ καλά το έργο μας. Είχαμε την υποστήριξη του Συμβουλίου και της Κομισιόν και πράγματι, όπως είπατε, σε ένα πολύ σύντομο χρονικό διάστημα μπορέσαμε να οργανώσουμε αυτή την αποστολή. Όπως είπατε, Πρόεδρε, εξετάσαμε και γενικά αλλά και λεπτομερή θέματα για να κάνουμε μια αναλυτική καταγραφή των στοιχείων από την πλευρά της υποεπιτροπής και διαπιστώσαμε ότι τα πιο σημαντικά θέματα είναι να μην ξαναεκραγεί η κατάσταση εξή, να μην ξαναρχίσει η σύραξη και να διατηρηθεί η σταθερότητα. Διαπιστώσαμε ορισμένε ελλείψεις όπου θα μπορούσαν τα πράγματα να είχαν εξελιχθεί καλύτερα. Πολλές φορές βέβαια όσοι κατηγορούν τι ευρωπαϊκές αποστολές προβάλλουν τα σφάλματα ή τι αδυναμίες. Αλλά εγώ πιστεύω πιστεύω ότι οι απόψεις μας πέρασαν, η ανταλλαγή αυτή των απόψεων ήταν πολύ σημαντική για να εκφραστούν οι θέσεις μας. Πιστεύω ότι η αποστολή αυτή είχε τεράστια επιτυχία, ιδίως μετά από την ε, συμφωνία που επιτεύχθηκε από το πρόεδρο Σαρκουζή να μπορέσουμε να προωθήσουμε και μη στρατιωτικό προσωπικό σε τόσο σύντομο χρονικό διάστημα. Ήταν το προσωπικό αυτό, τα στελέχη μας δηλαδή, λίαν, ε, συμπεριφέρθηκαν πολύ ε, επαγγελματικά, πολύ αποτελεσματικά και η Γεωργία ε, συμφώνησε να συνεργαστεί παραδείγματος χάρη στην ταυτοποίηση ε, στολών ε, και στη διαφοροποίηση στολών στρατιωτικού και μη στρατιωτικού προσωπικού ή στελεχών. Το μεγάλο πρόβλημα είναι βεβαίως η Νότια Ασετία και η θέση των Ρώσων εκεί, δεδομένου ότι δεν επέτρεψαν την επίσκεψή μας στην άλλη πλευρά των σύνορων. Επίσης η Απχαζία ε, σε αυτές τις δύο επαρχίες όπως είπαμε δεν μπορέσαμε να πάμε και διαπιστώσαμε στα σύνορα με την Νότια Οσετία επειδή δεν υπάρχουν επίσημες επαφές διαπιστώσαμε έτσι μια περίεργη ιεροτελεστία όπου υπάρχει μια ουδέτερη ζώνη τρεις προχωρούν από τη μία πλευρά και περιμένουν εν συνεχεία οι, νότιοι, οι, άνθρωποι από τη νότια Οσετία προχωρούν και αυτή στην νεκρή ζώνη και γίνεται μια κουβέντα σε αυτή την μια ανταλλαγή απόψε να θέλει σε αυτή την ε, νεκρή ζώνη από τη μία πλευρά υπάρχει ένα ρωσικό φυλάκιο και ένα ρώσικο τάγκ και από την άλλη πλευρά και, και ε, επίσης στους ε, κοντινούς λόφους μια έντονη στρατιωτική παρουσία των Ρώσων. Ε, περίεργη λοιπόν, πολύ το θέατρο του παραλόγου όπου εμείς άοπλοι αναγκαστήκαμε να μπούμε σε μια νεκρή ζώνη περιδρυγισμένη από όλο αυτό τον, τον οπλισμό και τις στρατιωτικές δυνάμεις των Ρώσων χωρίς να μπορούμε να περάσουμε, να προχωρήσουμε μέσα στο, στην Νότια Ισοτία. Ένα άλλο ε, θέμα είναι η ο σύνδεσμος, η επαφή με, τον σύνδεσμο από την πλευρά του ΟΗΕ ε, και το, της αποστολής του ΟΗΕ. Δηλαδή ο ξεματούχος σύνδεσμος ε, ποιος είναι, πώς θα διοργανώσουμε αυτή την επαφή η οποία δεν υπήρχε προηγουμένως μεταξύ ημών και το, του ΟΗΕ και αυτή η έλλειψη αξιωματούχου συνδέσμου ήταν πολύ απογοητευτική για τους ε, εργαζόμενους, για, για τους ανθρώπους που είναι εκεί. Ε, πιστεύω ότι ο ΙΕ πρέπει να παρακολουθήσει την κατάσταση εκεί και θέλει να το κάνει. Είναι ε, πολύ σημαντικό και για την υποστήριξη της Κομισιόν σε όλες αυτές τις δράσεις. Ε, οι προμήθειες επίσης ε, είναι δύσκολες για το προσωπικό μας σε αυτή την περιοχή, προμήθεια των απαραίτητων μέσων και υλικών. Ε, εμείς πήγαμε στην αποστολή αυτή χωρίς μια συγκεκριμένη ημερήσια διάταξη, γι' αυτό ακριβώς και δεν παρουσιάσουμε συγκεκριμένες προτάσεις στην υποπιτροπή είπαμε ότι θα ζητήσουμε να γίνουν περαιτέρω συζητήσεις και ανταλλαγές απόψε στο μέλλον. Δεν υπάρχει όμως καμία αμφιβολία ότι η σταθερότητα υπάρχει, έχει επιβληθεί, υπάρχει κατάπαυση πυρός ε, και όποιοι πυροβολισμοί ακούγονται είναι μάλλον από στρατιώτες ή πολίτες στην επικράτεια της Νότιας Οσετίας και δεν είναι ένοπλοι, ένοπλες σειράξεις. δεν υπάρχει καμία εγγύηση ότι δεν ξα, ξανασημειωθεί η σύραξη κάποια στιγμή Υπήρχε μάλιστα και μια συνέντευξη στην εφημερίδα ότι, που έλεγε ότι οι Ρώσοι θα αποτελειώσουν το έργο τους αυτό το καλοκαίρι και αναπόφευκτα θα δημιουργηθεί και μια άλλη σύραξη. Αλλά αυτά είναι μελλοντικά και αβέβαια και εικασίες. Εν πάση περιπτώσει, στα σύνορα επικρατεί σταθερότητα και το επιχείρημα που στηρίζει τη συνέχιση της αποστολή είναι το επιχείρημα της αναχέτης, της, ε, της, του να αποτρέψουμε ε, την μια νέα σύραξη. Είναι μια αποστολή αποτροπής. Έτσι ώστε εάν υπάρξει ένα προκλητικό επεισόδιο να μπορούν να, προληφ... να επιβληθούν, να γίνουν προληπτικές ενέργειες ώστε να μην ξανα ξανακαεί ε, η περιοχή, να, μην ξαναρχίσει λοιπόν η ένοπλη σύραξη. Ε, πιστεύω ότι ακριβώς αυτός ο ε, αποτρεπτικός ρόλος είναι ο βασικός ρόλος της αποστολής και ο άλλος ρόλος είναι επειδή οι Ρώσοι έχουν βέτο και στον ΟΗΕ ε, το οποίο βέτο θα το προβάλλουν τον Ιούνιο όταν λήξει η εντολή της αποστολής του ΟΗΕ το Σεπτέμβριο δεν θα θέλουν να επαναληφθεί θα προβάλλουν βέτο σε τυχόν πρόταση επανάληψης ή συνέχισης γι' αυτό μου είπαν ότι είναι πολύ σημαντικό όχι ποιος κάνει τη δουλειά σωστά εκεί επί τόπου, αλλά να γίνει η δουλειά σωστή, ό,τι χρειάζεται δηλαδή να γίνει. Τώρα από ποιον δεν έχει τόση σημασία όσο το αποτέλεσμα. Επισκεφθήκαμε και στα τόπεδα για τους εσωτερικά εκτοπισμένους και είδαμε πόσο γρήγορα στήθηκαν πρόχειρες ε, μονάδες στέγασης, πρόχειρες κατοικίες ή τέλος πάντων ε, κινητές μονάδες στέγασης Συναντήσαμε και έναν 94χρονο ο οποίος είχε πολεμήσει στον Ερυθρό στρατό στο Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο και ο οποίος αναγκάστηκε να φύγει ως πρόσφυγας από την Νότια Ισοτία και μας είπε με δάκρυα στα μάτια ότι δεν πίστευα ποτέ θα ξαναγίνω πρόσφυγας 94 μου χρόνια γι' αυτό ε, μετά από αυτά τα οποία που συνέβησαν. Βλέπετε λοιπόν ότι εσωτερικά εκτοπισμένη είναι ένα πολύ σημαντικό πρόβλημα και είναι αποτελεί και μια πολύ σοβαρή πτυχή των δράσεων της αποστολής να, να, να φροντίσει αυτούς τους ανθρώπους. πολλοί, πολλούς ε, πολίτες που συναντήσαμε εκεί ήταν ενθουσιώδεις και υποστήριζαν 100% τις προσπάθειες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και γι' αυτό πιστεύω ότι θα πρέπει να συνεχιστεί αυτή η αποστολή επίσης λαμβάνοντας υπόψη πόσο σημαντική είναι η γεωργία για τις ενεργειακές ε, προμήθειες στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Θέλω να καταλήξω με ένα πολύ θετικό πνεύμα και πρέπει να πούμε ότι ήταν μία, επιτέλους, μία πάρα πολύ επιτυχής ευρωπαϊκή αποστολή αυτή που θέτει ένα παράδειγμα, παραδειγματική δηλαδή και για άλλες αποστολές στο μέλλον παρόμοιες. Μικρόφωνο παρακαλούμε, ε, δεν ακούμε δυστυχώς. Ωραία. Κοιτάξτε, επειδή αναφερόμεθα στην επόμενη κοινοβουλευτική θητεία, θέλω να κάνω δύο παρατηρήσεις. Ε, το ένα θέμα το έφυξε η Πρόεδρος. Βεβαίως ε, σε αυτήν την ε, περιοχή δεν είναι σίγουρο κατά πόσον η Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει να διαδεχθεί μια αποστολή των ΗΠΑ Εθνών. Κατ' ουσίαν χρειαζόμαστε ένα όργανο όπου θα εκπροσωπούνται και οι Ρώσοι. Το δεύτερο, και το λέω αυτό ως εισηγήτρια για τα όργανα σταθερότητας, γιατί ο συνάδελφος μίλησε για αυτά και θέλω να του πω ότι κοιτάξτε το όργανο σταθερότητας αφορά τη γεωργία και από την άλλη αποδεσμεύονται κονδύλια έτσι ώστε να ανεγερθούν αυτές οι κατοικίες για τους εκτοπιστέντες. Προσπάθησα ε, να παρακαλώ στην Κομισιό να μας πει τι ακριβώς ε, σημαίνει αυτό. Μήπως είναι επικίνδυνο ο εθνικός διωγμός ή το δικαίωμα παλινόστησης των προσφύγων Ίσως με το να ε, δημιουργηθούν αυτά, αυτοί οι πρόσκαιροι ε, καταπλησμοί, αυτές οι πρόσκαιρες κατοικίες ε, ουδέν μονιμότερων του προσωρινού και τελικά μπορεί να παραμείνουν εκεί για πάντα και να τους εμποδίσει τους πρόσφυγες να επιστρέψουν στις αιστείες τους. Θεωρώ λοιπόν ότι αυτά τα κονδύλια ε, για την σταθερότητα στο μέλλον θα πρέπει κανείς να τα εξετάσει πολύ προσεκτικά γιατί σε τελική ανάλυση το όργανο σταθερότητας δεν έχει καμία σχέση με όλα αυτά. Πρόεδρος, ε, νομίζω ότι το ερώτημα είναι σωστό. Θα ήθελα να ευχαριστήσω τον συνάδελφο για την έκθεσή του και θέλω να του πω ότι ε, συμφωνώ και επαυξάνω. Η επίσκεψη που κάναμε στους εκτοπιστέντες ε, με εντυπωσίασε. Έχουμε, επισκεφθήκαμε δύο καταβλισμούς. Αυτούς οι οποίοι έφυγαν μετά την κατάρρευση της Σοβιετικής Ένωσης και εκείνους που διέφυγαν τώρα πρόσφατα. Κάναμε λοιπόν μία επίσκεψη ε, σε ένα καταβλισμό ε, προσφύγων ε, σε μια πολυκατοικία ήταν αυτή κατ' ουσίαν όπου οι εκδιοχθέντες ζουν εκεί υπό άθλιες συνθήκες εδώ και δέκα χρόνια. Ζουν εκεί και περιμένουν να επανέλθουν και το επιθυμούν αυτό διακαώς. Πρέπει όμως να πούμε ότι οι συνθήκες διαβίωσης των ανθρώπων αυτών είναι παντελώς απαξιωτικές. Και από την άλλη έχουμε αυτά τα σπίτια που χτίστηκαν πρόσφατα και εκεί ο στόχος ήταν να υπάρχουν ε, καταρχήν ε, δυνατότητες ε, διαμονής για αυτές τις 35.000 πρόσφυγες. Μιλάμε αυτές είναι σειρές, ατέλειωτες σειρές σπιτιών για οικογένειες όπου έχει κάνει την εντύπωση όταν τα έχει δει ας πούμε δεν υπάρχει εκεί καμία δυνατότητα αγοράς δεν υπάρχουν καταστήματα ε, δεν υπάρχει κανένα κέντρο για τα σπίτια είναι μια ατέλειωτη σειρά κατοικιών όπου το χειμώνα βέβαια επιβίωσαν οι άνθρωποι αυτοί. Δεν μπορώ να πω ότι αυτές οι κατοικίες είναι ελκυστικές έτσι ώστε να ε, πείσουν κάποιον να μείνει εκεί περισσότερο από ότι είναι απολύτως απαραίτητο. Γι' αυτό λοιπόν πράγματι είναι σωστό το να ε, χρησιμοποιηθούν εκεί και κονδύλια ε, σταθερότητος. Προφανώς η παραμονή εκεί δεν έχει προγραμματιστεί για το Δίνεκες. Κανείς δεν θέλει να μείνει εκεί για πάντα. Αλλά σας λέω, ήταν ε, βραχυπρόθεσμα απαραίτητο οι άνθρωποι να ε, μπορέσουν να περάσουν το χειμώνα. Και αυτό κοιτίζει το εξή ερώτημα. Κατά πόσον σε αυτή την κοινοβουλευτική θητεία θέλουμε να τοποθετηθούμε επί του θέματος ως ε, κοινοβούλιο ή να γίνει στην επόμενη. Εγώ νομίζω ότι η άποψη όσων συμμετείχαν στην αποστολή είναι ότι αν τελικά αυτό το θέμα, αν επαληφθεί ότι το θέμα δεν θα συνεχιστεί, τότε είναι ευθύνη της Ευρωπαϊκής Ένωσης να προγραμματίσει την παρέμβασή της για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα. Αυτό είναι το συμπέρασμα που εξάγω εγώ. Πρέπει λοιπόν να έχουμε κατά νου το εξής. Έχουμε λοιπόν τον προβληματισμό Γεωργία ΝΑΤΟ, Γεωργία Ευρωπαϊκή Ένωση ή αν θέλετε το ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση λίγο πολύ αποσύρεται από αυτή τη σύγκρουση και νομίζω ότι αυτό είναι ένα θέμα το οποίο θα πρέπει κανείς να το λάβει υπόψη του πριν ε, καταλήξει σε τελεσίδικη απόφαση. Νομίζω ότι μπορούμε να το κλείσουμε τώρα το θέμα και Πάμε τώρα έγκαιρα στην ώρα μας με το εργαστήριο κατάλοιπα πολέμου και ρήπανση της θάλασσας. Θα συνεχίσω στα αγγλικά. Σας καλωσορίζω λοιπόν σε αυτό το εργαστήριο που έχει σχέση με τη ρήπανση της ε, θάλασσας που προκαλείται από τα κατάλοιπα πολέμου. Αυτό έχει προβλεφθεί για να αξιολογήσουμε ε, της, ε, την καταστροφή που έχει προκύψει μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο που ε, έπληξε την Ευρώπη. Στόχος μας είναι να δούμε τι ακριβώς ποιες είναι οι επιπτώσεις της κατασκευής του North Stream προτείνεται η διαδρομή να περάσει και μέσα από τη Βαλτική θάλασσα. Ο αγωγός αυτός ε, θα μπορούσε να έρθει σε επαφή με τα κατάλοιπα εκεί των πυρομαχικών. Ε, χαιρετίζουμε τον ε, πρόεδρο της Λιθουανίας στην Ολλανδία, ο οποίος ήρθε ειδικά για αυτή τη συνάντηση. Σας καλωσορίζουμε λοιπόν κοντά μας. Πρέσβης εννοείται. Είναι λοιπόν το εργαστήριο αυτό το οποίο ε, θα ξεκινήσει με την παρουσίαση του κυρίου Τζον Χάρτ ο οποίος ε, εργάζεται για το Διεθνές Ινστιτούτο Ερευνών της Στοκχόλμης ε, για την Ειρήνη, πρόγραμμα χημικού και βιολογικού πολέμου. Έχει 15 λεπτά στη διάθεσή του για να μας παρουσιάσει τα αποτελέσματα της μελέτης και κατόπιν θα ακολουθήσει ο κύριος Τζέφρι Οσπον ο οποίος εργάζεται για τον, το, στο τμήμα επαλήθευσης του Οργανισμού για την Απαγόρευση των Χημικών Όπλων στη Χάγη και κατόπιν ο κ. Μακ Κοχ, ερευνητής ε, στο Πανεπιστήμιο του Λούνεμπουργκ. Ο καθένας έχει περίπου 10 ε, λεπτά για να παρουσιάσει την ομιλία του. Και κατόπιν θα ακολουθήσει η συζήτηση από τα μέλη και από τους εμπειρογνώμονες. Ε, τους καλωσορίζω όλους θερμά και δίνω το λόγο στον πρώτο μιλητή.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 Ευχαριστώ Πρόεδρε. Θα ήθελα να ευχαριστήσω τους δύο για τη δυνατότητα που μου δίνουν να παρουσιάσω σήμερα το έγγραφό μου. Να ευχαριστήσω επίσης και τον Δ. Κουέλ και όλους τους υπόλοιπους που κατέστησαν δυνατή αυτή την παρουσίαση. Θα ήθελα να ευχαριστήσω για την ευκαιρία που μου δώσατε να έρθουν και δύο εξωτερικοί συνεργάτες ε, προκειμένου να σχολιάσουν την παρουσίαση. Πολύ σύντομα λοιπόν θα σας δείξω μερικές διαφάνειες. Μυστικώς οι διερμηνείς δεν βλέπουν τις διαφάνειες. Αν θέλετε κάποια αντίγραφα θα μπορούσα να σας αφήσω με τις διαφάνειες ή μπορείτε να μου στείλετε και ένα mail, εάν ενδιαφερόσαστε. Εν συντομία λοιπόν θα αναφερθώ σε κάποιες από αυτές τις ε, διαφάνειες. Να ξεκινήσω λέγοντας ότι υπάρχουν μεγάλες ποσότητες ε, όπλων που παράγονται παγκοσμίω και, και έχουν αποθηκευτεί σε διάφορα σημεία ειδικά μετά τον πρώτο και τον δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο υπήρξαν πάρα πολλά πολεμοφόδια τα οποία είχαν αποθήκευθεί και συνήθως αυτή η αποθήκευση γινόταν είτε με πόντιση στις θάλασσες είτε αποθήκευση στα έδαφος. Κάθε χρόνο, κάθε μήνα ανακαλύπτουμε πολεμοφόδια και είναι δύσκολο να πούμε πως ε, πολεμοπόδια έχουν ποντιστεί στην Βαλτική θάλασσα. Ε, γίνονται ε, συχνά ανακαλύψεις ακόμα και βυθισμένων πλοίων. Σε ό,τι φορά τη Βαλτική θάλασσα, η περισσότερη δουλειά που έχει γίνει, γίνει στο πλαίσιο της Συμφωνίας του 1992 για την προστασία του θαλάσσιου περιβάλλοντος στην Βαλτική. Ζητά συγγνώμη ο αγορητής επειδή διαβάζει πολύ γρήγορα και υπάρχει η Επιτροπή του Ελσίνκη που ασχολείται το 99 κατεβήξαν προσπάθειε προκειμένου να μάθουμε περισσότερο για την πόντιση πυρομαχικών στην Βαλτική. Ένα από τα μέσα που έχουμε είναι ο υπολογισμό σε τόνους. 3.500 τόνοι πυρομαχικών υπολογιστήρων ότι έχουν ποντιστεί στην Βαλτική. Υπάρχει μια άλλη εκτίμηση 168.000 τόνων μόνο και μόνο στην περιοχή του Σκαγεράκη. Uh, I think I'll skip a few of these other things. Τώρα θα σας δείξω μερικές φωτογραφίες. Νομίζω η φωτογραφία στα πάνω αριστερά. Πρόκειται για ένα πλοίο. Μιλάμε για μια επιχείρηση του 1916. Δεξιά Νομίζω πως υπάρχει κάποιο εμπορευμένο κυβότιο, αλλά υπάρχει δίπλα μου ένας εμπειρογνώμος που τα ξέρει καλύτερα και κάτω υπάρχουν φωτογραφίες από την Βαλτική. Πρόκειται για φωτογραφίες που προχωρούνται από ένα εγχειρίδιο το οποίο είχε, είχε στόχο να βοηθήσει τους ψαράδες να ανοιχνεύουν πυρομαχικά. Υπάρχουν και τορπίλες ε, βόμβες ε, βλέπετε κάτω δεξιά νάρκες εδώ βλέπετε έναν άλλο χάρτη που προέρχεται από μια έκθεση και δείχνει τις περιοχές όπου ε, βρίσκονται χημικά όπλα Αλλά φυσικά οι μεγαλύτερες ποσότητες των πυρομαχικών που έχουν ποντιστεί, έχουν ταφεί, είναι συμβατικά όπλα και πυρομαχικά. Βλέπετε εδώ κάποιες άλλες δραστηριότητες, οποίες ε, θα αποφύγω να σχολιάσω. Όλα αυτά προέρχονται από πληροφορίες που έχουμε λάβει σε, από κάποια έγγραφα δεν θα σας κουράσω περαιτέρω με αυτές τις λεπτομέρειες. Και εδώ βλέπετε μια άλλη διαφάνεια που αφορά γενικές παρατηρήσεις για τα χαρακτηριστικά των πυρομαχικών, συμβατικών αλλά και χημικών. Για αυτή τη διαφάνεια Θα ήθελα να πω ότι συμμετέχουν διάφοροι εμπλεκόμενοι. Ορισμένοι εργάζονται στο πρόγραμμα πλαίσιο, το έκτο πρόγραμμα πλαίσιο, το οποίο αφορά έρευνες στην Βαλτική και εφαρμόζουν μια συγκεκριμένη προσέγγιση προκειμένου να εντοπίσουν τα πυρομαχικά αυτά. υπάρχουν όμως και διάφορες ομάδες ε, ανθρώπων που ασχολούνται με το ψάρεμα που όμως ε, παράλληλα κάνουν αυτές τις έρευνες. Υπάρχουν και κάποιες βάσεις δεδομένων για λόγους αναζήτησης αρχαιοτήτων κλπ. Υπάρχουν λοιπόν βλέπετε πολλές ε, πολλοί τρόποι για να ενημερωθούμε σχετικά με την ε, ύπαρξη πονισμένων πυρομαχικών ε, Αυτά είναι, είναι κάποιες γενικές πληροφορίες περιβαλλοντικής φύσης και θα ήθελα, θα πρέπει όμως να παραμείνω μέσα στο χρόνο που μου δώσατε, άρα δεν μπορώ να σας πω και πάρα πολλά. Να αναφέρω τώρα κάποια θέματα που αφορούν την ανθρώπινη υγεία. Θα πρέπει να κάνουμε διάκριση ανάμεσα στι διάφορες μορφές ε, τοξικότητας υπάρχουν ε, κάποιοι τρόποι διαβάθμισης ε, της τοξικότητας. Ορισμένες φορές δυστυχώς δημιουργείται κάποια σύγχυση για τα επίπεδα τοξικότητας και είναι δύσκολο να εφαρμοστούν η διαβάθμιση αυτή για τα διάφορα είδη ζώων. Εάν Μάλλον αυτό το οποίο αναφέρεται συχνά είναι η τεχνητή τοξικότητα. Κάτι το οποίο παράγεται από τον άνθρωπο μπορεί να είναι περισσότερο τοξικό Επίσης αυτό που έχει σημασία νομίζω είναι ότι πρέπει να έχουμε κατά νου ε, την διάλυση και την ε, διάχυση. Ε, δεν έχω εδώ ακριβείς υπολογισμούς, αλλά αυτό που παίζει ρόλο είναι ότι όταν ένας διαλύτης έχει διαχυθεί στη θάλασσα, βεβαίως διαχέεται και ένα άλλο θέμα σημαντικό είναι ότι όταν υπάρχει ο κίνδυνος, ε, υπάρχει ο κίνδυνος ε, μόλυνσης όταν καταστρέφει κανείς μία χωματερή. Νομίζω λοιπόν ότι το διοξίδιο του θείου είναι ένας, ε, μια ουσία ε, η οποία προκαλεί εκρήξεις και υδρογονώνεται πολύ εύκολα όταν η θερμοκρασία είναι πολύ υψηλή εκεί πρέπει να γνωρίζουμε ότι υπάρχει κίνδυνο στο εσωτερικό ε, να παραμείνει με τη μορφή του εξόδους Ένα άλλο θέμα... Ένα άλλο θέμα που είναι ενδιαφέρον είναι η μόλυνση, η ρήπανση με αρσένιο. Ε, δεν θα ήθελα εδώ να μπω σε λεπτομέρειες. Ε, και κατόπιν υπάρχει και μια άλλη κατηγορία ε, των ε, συμβατικών ε, πυρομαχικών ε, που και αυτά έχουν χρησιμοποιηθεί και μπορούν να προκαλέσουν σημαντική ρήπανση. Δεν θα ήθελα να αναφερθώ γιατί έχω κάποια συγκεκριμένα στοιχεία για την τοξικότητα όλων αυτών των ουσιών αλλά δεν θα μπω σε λεπτομέρειες, θα ήθελα να περάσω στα συμπεράσματα. Υπάρχει λοιπόν εδώ, ε, βλέπετε, ένας κατάλογος που δεν θέλω να σας τον διαβάσω, όμως υπάρχει το δεύτερο σημείο που αφορά τη σημασία των τοξικολογικών ε, ερευνών και των μηχανισμών αναφοράς. Αν σκεφτεί κανείς τους μελλοντικούς τομείς ε, δραστηριοτήτων, θα διαπιστώσει ότι υπάρχουν διάφοροι μηχανισμοί που υφίστανται έτσι ώστε συστηματικά να συγκεντρωθούν, ε, να επικαιροποιηθούν και να αναφερθούν τα τοξικολογικά στοιχεία. Αυτό που μπορεί κανείς να δει είναι η ε, εφαρμογή της καταχώρησης, της αξιολόγησης ε, και του περιορισμού των χημικών ουσιών του περίφημου ακτικόλεξου REACH. Υπάρχει και ο οργανισμός που ελέγχει όλα αυτά και που άρχισε να συλλέγει πληροφορίες ε, σε καθαρά προαιρετική βάση. Τούτο συνέβη πέρυσι. Ε, πάνω από 65.000 εταιρείε έχουν καταθέσει δύο έχουν καταθέσει πάρα πολλές ε, αιτήσει για καταχώρηση. Υπάρχει η τράπεζα δεδομένων, Uniform Chemical, είναι μια τράπεζα δεδομένων ε, που περιλαμβάνει ε, τα σχετικά στοιχεία. Αυτό που θέλουμε να πούμε είναι ότι για λόγους ασφαλείας υπάρχει ε, μια σειρά νέων απαιτήσεων με στόχο να καταδειχθεί ότι μια χημική ουσία δεν προκαλεί απαραίτητα ζημιά. Είναι σημαντικό αυτό και δεν πρέπει να περιμένουμε απαραίτητα ώστε να προκύψει μια πληροφορία ότι πράγματι μια χημική ουσία προκαλεί ρήπανση. Μπορεί να είναι προβληματική η επιλογή κάποιων ε, τεχνολογικών εφαρμογών όταν υπάρχει ε, πόντιση ε, πυρομαχικών Πολλοί διαφωνούν με την καύση, κυρίως όταν αυτή γίνεται ε, σε χερσαία βάση. Ένα βασικό ερώτημα είναι κατά πόσον θα πρέπει κανείς να κάνει κάτι να μην κάνει απολύτως τίποτα. Εγώ όμως νομίζω ότι η επικρατούσα άποψη και αυτό το υποστηρίζουν και εμπειρογνώμονες, απορρευνητικά Ινστιτούτα και επιστήμονες ότι λόγω του ότι δεν υπάρχουν αποχρόντες λόγοι που να οδηγούν στο ότι πρέπει να γίνει κάτι καλύτερα τα πυρομαχικά να παραμείνουν εκεί που έχουν ποντιστεί έχουν ποντιστεί βαθιά στη γη, ε, τα ποσοστά διάβρωσης τους ε, είναι ανεκτά. Ε, υπάρχουν μελέτες που προσπαθούν να συγκεντρώσουν καλύτερα στοιχεία για τη διάβρωση, αλλά και σε μεμονωμένες περιπορώ ότι είναι καλύτερα να αφήσει κανείς εκεί το πυρομαχικό ακόμα και αν είναι απόλυτα διαβρωμένο. Ε, ορισμένα πυρομαχικά εγκλωβίζονται μέσα σε κομμάτια από μπετόν. Εκείνο που είναι απαραίτητο είναι να συνεχιστεί η αξιολόγηση έτσι ώστε να υπάρχει καλύτερη κατανόηση του επίπεδου ρήπανσης της Βαλτικής γενικότερα. Εξάλλου είναι όλο και πιο δυνατό ε, να συγκεντρώσει κανείς τα δεδομένα τα οποία αποκτά μέσω διαφόρων μηχανισμών. Πληροφορίες δηλαδή που παράγονται από ανθρώπους που θέλουν να διατηρήσουν ε, κάποια ναυάγια ή ε, Ας μην ξεχνάμε ότι η Βαλτική θάλασσα είναι αρκετά ρηχή και εκεί διαφυλάσσεται πάρα πολύ καλά η ιστορία του κόσμου. Νομίζω ότι υπάρχει μεγάλο περιθώριο να γίνουν και άλλες έρευνες χρησιμοποιώντας ε, πηγές εκτός ε, της αγγλικής που δεν είναι στην αγγλική γλώσσα. Όλα τα υπόλοιπα στοιχεία μπορείτε να διαβάσετε τη διαφάνειά μου. Θέλω να καταλήξω στο εξή. Όποια προσέγγιση και αν επιλέξει κανεί να κάνει ή να μην κάνει κάτι, είτε αυτό σημαίνει την ανάκτηση των πυρομαχικών με διαφορετικού τρόπου ή την εφαρμογή νέων ε, καθεστώτων και πρωτοκόλων ελέγχου, σε τελική ανάλυση εκείνο που παίζει ρόλο είναι ότι η τεχνική λύση θα πρέπει να είναι και εφαρμόσιμη. Αν δηλαδή υπάρχει κάποιο χάσμα ανάμεσα στην ανάκτηση των συμβατικών ή των χημικών πυρομαχικών και της ε, πολιτικής ή της ε, ε, πολιτικής πίστης, κοινής γνώμης, οποιοδήποτε τέτοιο χάσμα θα πρέπει να αντιμετωπιστεί και οποιαδήποτε προσέγγιση επιλογή θα πρέπει να χαρακτηρίζεται από ισορροπία και σύνεση. Βεβαίως αυτό πάλι είναι καθαρά υποκειμενικό. Εν πάση περιπτώσει, ε, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Ο επόμενος ομιλητής μα είναι ο κύριος Τζέφρι Όσμπορν. Uh, ευχαριστώ Πρόεδρε που μας δίνετε την ευκαιρία να συμμετάσχουμε σε αυτό το φόρουμ και ευχαριστώ και όλους που συνεργάστηκαν για την προετοιμασία. Υπάρχουν ορισμένες ε, εικόνες, ορισμένες διαφάνειες που μπορεί να σας βοηθήσουν Είμαι ο Τζέφρι Osborne από τον Οργανισμό για την Απαγόρευση των Χημικών Όπλων και εργάζομαι στο τμήμα υπαλήθευσης και ιδίως ε, για τα χημικά και βιολογικά που, που, που κατασκευάστηκαν πριν από το 1946. Η σύμβαση για τα χημικά είναι μια διεθνή ε, σύμβαση για την επαλήθευση των χημικών όπλων διεθνώς ε, και για να βοηθήσει και στον τομέα της, ε, της χημίας και για όλους τους συναφείς τομείς για την κατασκευή των όπλων. Ο οργανισμός αυτός, ο ΑΧΟΒ, εδρεύει στη Χάγη, στις κάτω χώρες. Όσον αφορά τώρα τα χημικά όπλα, παρακολουθούμε στενά τη δήλωση, αποθήκευση και καταστροφή και των χημικών όπλων αλλά και των εγκαταστάσεων παραγωγής. Έχουμε μία, ε, ένα, μία μονάδα αποστρατικοποίησης η οποία είναι υπεύθυνη για να προκολουθήσει την καταστροφή των χημικών όπλων. Αυτή η μονάδα αποστρατικοποίησης εμπίπτει ε, στην ε, λειτουργεί πάνω από την, κάτω από την εποπτεία του οργανισμού μας, ο ΑΧΟ. Ο οργανισμός, ο ΑΧΟ, ασχολείται επίσης με την ανάκτηση των χημικών που έχουν ποντιστεί και καταγράφουμε τις διαφορετικές ε, θέσεις ε, των κρατών μελών μας όσον αφορά την ανάκτηση των χημικών στοιχείων αυτών από ποντισμένα όπλα η γραμματεία μας λειτουργεί με αυστηρές τεχνικές προδιαγραφές για την επαλήθευση, αποθήκευση και καταστροφή αυτών των όπλων ε, κάτω από το καταστατικό του οργανισμού μας, του οργανισμού απαγόρευσης. Θα ήθελα να σας εξηγήσω λίγο τις ε, απαιτήσεις του ΟΑΧ όσον αφορά την πόντιση χημικών όπλων. Μία απέτηση κλειδί είναι ότι όποιος θέλει να ποντίσει χημικά όπλα πρέπει να τα δηλώσει και πρέπει να δηλωθούν αυτά τα χημικά όπλα εάν και όπου αποθηκεύονται στην επικράτεια του, αυτού, αυτού που δηλώνει. Τα όπλα αυτά τα χημικά που κατασκευάστηκαν πριν από το 1946 πρέπει να δηλωθούν Κάθε μέλος που έχει συνυπογράψει τον οργανισμό μας πρέπει να δηλώσει αν στην επικράτειά του έχει αυτά τα όπλα, τα παλιά, τα χημικά, έτσι ώστε εμείς να μπορούμε να επισκεφθούμε και να τα επαληθεύσουμε. Επίσης, θα πρέπει να δηλώσει αν υπάρχουν εγκαταλειμμένα όπλα. Πρέπει δηλαδή να μας δώσει όλες τις πληροφορίες για τυχόν παπαλαιωμένα όπλα τα οποία περιέχουν χημικά για να μπορούμε εμείς να εκτελέσουμε τον ρόλο της επαλήθευσης πριν ε, από το, τον Ιανουάριο 1997 ή η πόντιση πριν από το 1985 δεν είναι υποχρεωτικό να δηλωθεί. Εάν όμως 77, 1977. Εάν όμως διαπιστώσουμε ότι υπάρχουν τέτοια όπλα θα πρέπει να δηλωθούν και να καταστραφούν σύμφωνα με τις όρους της συνθήκης. Μόνο ένα κράτος μέλος έχει δώσει πληροφορίες για αυτά τα πιο σύγχρονα χημικά όπλα που έχουν ποντιστεί επί τη βάση ε, των διατάξεων για το 1977 όπου δεν προβλέπεται υποχρεωτική δήλωση. Τα περισσότερα όπλα με χημικά, ε, χημικά έχουν, ε, έχουν ε, σε χωματερές στο έδαφος δηλαδή, όχι στη θάλασσα. Και η ανάκτηση και η ουδετεροποίηση είναι πιο δύσκολη και πολύ πιο επικίνδυνη. Κανένα από τα κράτη-μέλη δεν έχει δηλώσει ότι έχει ποντίσει επικίνδυνα χημικά όπλα. Ναι. Ε... Αυτά ήταν χημικά όπλα, όσα όπλα καταγράφτηκαν ότι βγήκαν από τη θάλασσα, από το βυθό της θάλασσας, ήταν όπλα τα οποία είχαν βυθιστεί κοντά στις παράκτιες περιοχές που δεν έπρεπε να έχει γίνει βεβαίως. Όμως δυστυχώς έχει επισημανθεί ότι αυτές οι περιπτώσεις υπάρχουν, έχουν καταγραφεί. Εν συνεχεία βεβαίως δηλώθηκαν και καταστράφηκαν τα όπλα αυτά βάσει με τη συνθήκη απαγόρευσης. Αυτό έχει συμβεί, το, φαινόμενο αυτό στην Ιταλία, στο Ηνωμένο Βασίλειο, που εξευράστηκαν δηλαδή χημικά όπλα στις ακτές, τι Ηνωμένε Πολιτείες και την Ιαπωνία. Έχουμε μια τεράστια εμπειρία και κανένας άλλος φορέας δεν έχει τόσο καλή εμπειρία και πλούσια εμπειρία όσο έχουμε εμείς για την ανάκτηση, εξουδετέρωση και επαλήθευση. Έχουμε εφαρμόσει μια ευέλικτη τακτική και αναγνωρίζουμε ότι κάθε κράτος έχει διαφορετικά προβλήματα, διαφορετικές δυνατότητες, διαφορετικούς πόρους, διαφορετική αντιμετώπιση. Κάθε Κάθε τοποθεσία την οποία διαπιστώνουμε είναι διαφορετική. Κάθε ανάκτηση είναι δύσκολη, είναι διαφορετική και πρέπει να, να γίνει με την, κατά το βέλτιστο τρόπο. Ο ΑΧΑ συνεργάζεται με τα κράτη-μέλη στην τεχνική βοήθεια, στην αναθεώρηση διαδικασιών και στην έγκριση ειδικών έκτακτων ε, διαδικασιών σε ορισμένες περιπτώσεις προσφέρουμε τεχνική βοήθεια επιτόπου για να δούμε αν τα, ποια είναι τα επικίνδυνα χημικά τα οποία περιέχονται στα όπλα ε, και γίνεται λοιπόν ε, μία επίσκεψη της ομάδας τεχνικής επαλήθευσης. Αυτή είναι μία διαφορετική από την κανονική επαλήθευση την οποία γίνεται από την άλλη διαδικασία. Είναι καθαρά τεχνική βοήθεια, τεχνική στήριξη. Οπότε, εν συνεχεία, η τεχνική ομάδα μπορεί να προχωρήσει ε, αφού αποφασίσει ποιος είναι ο καλύτερος τρόπος για να εξουδετερευθούν τα χημικά όπλα. Αυτό έχει γίνει, τεχνική υποστήριξη δηλαδή, ήδη στην Αιθιοπία, στη Βιετνάμ και στο Παναμά. Επίσης προσφέραμε τεχνική βοήθεια στην Ιταλία πριν από δύο χρόνια, όταν ανακάλυψαν ένα τεράστιο οπλοστάσιο, συμβατικό βασικά, σε μία συγκεκριμένη τοποθεσία την πρώτη ε, εβδομάδα πάνω από 600 χημικά όπλα εντοπίστηκαν, διαχωρίστηκαν και καταγράφτηκαν και συνεχεία καταστράφηκαν από την Ιταλία. Η γραμματεία του οργανισμού έχει ε, ε, αλλάξει τους κανονισμούς για να μπορέσει να βοηθήσει την Ιαπωνία στην ανάκτηση, επαλήθευση και καταστροφή χημικών όπλων πρώτους 1946 κατά τρόπο που, που, που να σέβεται τις διατάξεις της ε, σύμβασης. Πρόσφατα είχαμε μία περίπτωση στην Αυστρία, όπου για πρώτη φορά μετακινήθηκαν ε, χημικά όπλα πρώτου 1946, κατασκευαστέντα δηλαδή, σε άλλες δύο γειτονικέ χώρες για καταστροφή όποτε διαπιστώνεται, όποτε βρίσκουμε, είτε στο έδαφος, ε, στη γη, είτε στη θάλασσα χημικά όπλα, η όλη διαδικασία εξουδετέρωσης, ανάκτησης και εξουδετέρωσης είναι πάρα πολύ δύσκολη. Από τη στιγμή όμως που ανακτώνται τα όπλα αυτά πρέπει να καταγραφούν, να πολιτευθούν και να καταστραφούν με το σωστό τρόπο. Βασικά ο μεγαλύτερος στόχος μας του οργανισμού ΑΧΟ είναι η καταστροφή των χημικών όπλων αυτών και η τεχνική γραμματεία όποτε της γίνει αναφορά για την ότι εντοπίστηκαν τέτοια όπλα είναι πάντοτε στη διάθεση της ε, χώρας η οποία κάνει τη δήλωση αυτή και οι διαδικασίες που εφαρμόζονται είναι πάντοτε διαφανείς και βασίζονται στην αλληλοενημέρωση με όλους τους ενδιαφερόμενους. Ό, όσοι δεν ξέρετε, βλέπετε εδώ στην διαφάνεια παραδείγματα από τις ε, δράσεις μας τι βρέθηκε, ε, τι απλοστάσια από βόμβες βρέθηκε πάνω σε αυτό το πλοίο. Περίπου 3.000 βόμβες εντοπίστηκαν πάνω στο πλοίο αυτό. Σας ευχαριστώ και ο επόμενος ομιλητής είναι ο κύριος Κόχ. καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Σας ευχαριστώ κύριε Von Βόγκο, ε, που με καλέσατε. Τα επόμενα 10-12 λεπτά θα ασχοληθώ με τη Βαλτική θάλασσα ε, και θα σας παρουσιάσω ένα κομμάτι της διατριβής μου που θα παρουσιάσω την επόμενη εβδομάδα στο Πανεπιστήμιο της Λούμπεκ. Λοιπόν, πρώτα απ' όλα μια εισαγωγή για, τον, ε, ε, για τα πυρομαχικά που έχουν βυθιστεί στην Βαλτική θάλασσα. Θα εξετάσουμε τον κίνδυνο ε, που συνεπάγονται την ανάγκη δράσης και θα καταλήξω μετά από 12 περίπου λεπτά. Πρώτα απ' όλα να πω ότι οι χωματερές κάτω από την επιφάνεια της θάλασσας ε, υπάρχουν σε ε, θάλασσες, σε μικρούς ποταμούς και ε, μικρές λίμνες. Πρέπει λοιπόν να διαχωρίζουμε ανάμεσα σε χημικά και συμβατικά όπλα γιατί και τα δύο έχουν ιδιαίτερα χαρακτηριστικά και οι κίνδυνοι που απορρέουν από τα χημικά όπλα είναι κατά κανόνα πολύ μεγαλύτεροι. Ε, τα χημικά ε, πυρομαχικά ε, πρόκειται κυρίως από το αχρησιμοποιητό οπλοστάσιο του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου και κυρίως λόγω του ότι την εποχή εκείνη δεν υπήρχε τεχνολογία για να καταστρεφούν αυτά τα πυρομαχικά. Ο ποντισμό στη θάλασσα έμοιαζε να είναι ο πιο αποτελεσματικός τρόπος για να ε, ξεφορτωθεί κανεί ένα εκατομμύριο συμβατικά όπλα μετά την ε, πάυση του πυρός ε, στη Γερμανία από το 45 μέχρι το 48 και την ε, ανάκληση της επιστράτευσης. Βλέπουμε λοιπόν ότι όσον αφορά την πόντιση λόγω του κόστους αποκλείστηκε η πόντιση στον Ατλαντικό. Η Βαλτική ήταν πιο βολική, πιο εύκολη λύση. Το βάθος είναι 10 ε, μέχρι 100 μέτρα και στο Σκάργακ ε, το βάθος είναι 600 μέτρα. Τα χημικά πυρομαχικά ε, ποντίστηκαν στο Σκάργακ στη Βαλτική θάλασσα. Τα συμβατικά πυρομαχικά ποντίστηκαν στη Βόρεια θάλασσα κοντά στην ακτή. Βλέπουμε λοιπόν εδώ τους ε, ειδικού ε, που καταστρέφουν τα όπλα αυτά, ε, τα σκεπάζουν με χώμα, μερικές φορές τα τοποθετούν σε σημεία ανοιχτής καύσης. Αυτό εδώ είναι με φωτογραφία του Σκάργακ όπου τα χημικά πυρομαχικά ήταν τοποθετημένα πάνω σε ρημουλκά και το άλλο που βλέπουμε είναι στο Bonhomme, εκεί η πόντιση έγινε από Γερμανούς εργάτες με το χέρι, ε, χωρίς ε, κανένα προστατευτικό εξάρτημα. Και γι' αυτό προέκυψαν και φρικαλαία ατυχήματα. Τώρα, τα σημεία πόντισης στη Βαλτική θάλασσα. Έχουμε συμβατικά, πυρομαχικά Έχουμε την περιοχή του Bay, την περιοχή του Σκάργακ, την ευρύτερη περιοχή. Αυτά είναι τα βασικά σημεία πόντισης. Έχουμε το Κάρτεγκαρτ, Γκότλαντ και το Μπονχόλμ. Το Μπόνχολμ είναι ε, το κυριότερο σημείο πόντισης. 180.000 τόνοι ε, χημικών και συμβατικών όπλων, αλλά κυρίως χημικών πυρομαχικών, ε, ποντίστηκαν στο Σκάργακ αποκινούμε 74 σκάφη. Έχουμε 32.000 τόνους ε, χημικών πυρομαχικών που ποντίστηκαν ανατολικά του Μπονχόλμ και επίσης 2.000 τόνους στο Κόνχαμ για τη Βαλτική ε, δεν έχουμε αξιόπιστα στοιχεία για συμβατικά ε, πυρομαχικά. Έχουμε όμως περίπου 100.000 πυρομαχικά που έχουν ποντιστεί κάτω από τις ε, γερμανικές ακτές. Επίσης έχουμε και ένα πολύ μεγάλο αριθμό ανεπίσημων σημείων πόντισης, χωματερών αν θέλετε, Έχω βρει πάρα πολλές εξ αυτών κατά τη διάρκεια της διατριβή μου. Αυτά έγιναν στα τέλη της δεκαετία του 80 ε, και έχουμε και ε, πυρομαχικά των ε, ελαφραίων, ελαφρών δυνάμεων που ποντίστηκαν μαζί με τα πυρομαχικά αυτά. Υπάρχει και μια φήμη ε, που αναφέρει ότι υπήρξαν και συνεργασίες για την πόντιση πυρομαχικών στη Βαλτική και υπάρχουν και διάφορες φήμοι για ε, βιολογικό υλικό το οποίο ενδεχομένως έχει ποντήσει η Ρωσία. Όσον αφορά αυτά τα χημικά πυρομαχικά Το μεγαλύτερο πρόβλημα που προκαλείται είναι το coconut effect, η επίδραση της καρύδας αν θέλετε, ανοίγει κατά κάποιον τρόπο το πυρομαχικό. Αυτά τα ε, πυρομαχικά ε, προστατεύονται ιδιαίτερα, ε, κυρίως κατά τη μεταφορά τους. Όσον αφορά τώρα τους κινδύνους ε, ενδεικτικά θα ήθελα να σας πω υπάρχει μεγάλη τοξικότητα σε περίπτωση άμεσης επαφής. Αυτό ε, το γνωρίζουμε από ψαράδες που ήρθαν σε επαφή με αυτά τα πυρομαχικά. Είχαμε 450 περιπτώσεις ατυχημάτων ε, με ψαράδες τα τελευταία 22 χρόνια. Έχουμε το πρόβλημα της χρόνιας τοξικότητας όταν ε, τα ε, πυρομαχικά είναι εμπλουτισμένα και κυρίως αυτά μπορούν να μπουν και στην τροφική αλυσίδα. Ε, αυτά προκαλούν καρκίνους και μεταλλάξεις. Υπάρχουν αυτοί οι κίνδυνοι. Εξάλλου είναι δυνατόν αυτά να δημιουργήσουν πρόβλημα και σε περίπτωση τρομοκρατίας έχουν ποντιστεί και λίγο έξω από το Βέλγιο πυρομαχικά σε βάθος 5 μέχρι 10 μέτρων. Ή είναι δυνατόν να κλείεται ε, ξαφνικά τοξικό της ε, γιατί ενδέχεται ένα πλοίο να προσκρούσει στο Σκάργκεκ ή ε, να προκληθούν αλυσιδωτές αντιδράσεις μέσω της αυτοανάφλεξης, αυτοέκρηξης. Και υπάρχει και η ε, διάβρωση που οδηγεί στο ότι δεν μπορεί κανείς να χειριστεί καλά αυτά τα πυρομαχικά και αυξάνεται κατά πολύ βεβαίως και η τοξικότητα τους. Η ανάγκη δράσης, το τι λοιπόν πρέπει να κάνουμε, έχουμε αφενός ε, όλο και μεγαλύτερη ανησυχία σχετικά με τα σημεία πόντισης ε, και το οικολογικό, τοξικολογικό δυναμικό το οποίο περικλείουν Έχουμε όλο και μεγαλύτερη πίεση ε, που βασίζεται στο ότι διαπιστώνεται διάβρωση και είναι όλο και πιο δύσκολο να χειριστεί κανείς τα πυρομαχικά αυτά εφόσον αποφασίσει να τα ανακτήσει. Και από την άλλη υπάρχει όλο και μεγαλύτερη ε, διαθεσιμότητα τεχνολογίες για να τα ανακτήσει κανείς ε, με ασφάλεια, με ρομπότ, ε, με σωστά μέτρα μεταφοράς, με θαλάμους, τους χάρη έκρηξης, ανάφλεξης αυτών των πυρομαχικών. Το συμπέρασμά μου είναι ότι δεν μπορεί κανείς να αποφύγει ε, τα προβλήματα τοξικότητας. Ε, η κατάσταση στη Βαλτική που πρέπει να αντιμετωπιστεί είναι ιδιαίτερη και δεν υπάρχει προηγούμενο. Το να μην δράσει κανείς τα επόμενα χρόνια αυτό σημαίνει ότι θα δημιουργηθούν ανεπίλητα προβλήματα που θα πλήξουν πάρα πολλές επόμενες γενναίες. Σας ευχαριστώ πολύ για την παρέμβασή Να δώσω το λόγο τώρα στον ε, Λιθουανό πρεσβευτή στην ε, Ολλανδία, εξχωρητά του Βοϊντάτας Βέρμπα. Ευχαριστώ Πρόεδρε, αξιότιμα μέλη του Κοινοβουλίου. Χαίρομαι που μου δίνετε αυτή την ευκαιρία να κάνω κάποιες παρατηρήσεις ε, από πλευράς Λιθουανίας σχετικά με την απαγόρευση, σύμφωνα με τη συμφωνία της Χάγης για την απαγόρευση χημικών όπλων. Τα πόντιση χημικών όπλων και πυρομαχικών είναι ένα ζήτημα που ανησυχεί και πολλούς και εξετάζει σε πολλά διεθνή φόρα. Το πρόβλημα έγινε στο ότι δεν υπάρχουν στοιχεία ε, σχετικά με το που έχουν πονηθεί, αυτά τα πυρομαχικά προκειμένου να περιορίσουμε τους κινδύνους για τους, το για τους ανθρώπους και για το περιβάλλον. Μέχρι τώρα δεν έχουμε ε, εκθέσεις ε, για το που βρίσκονται αυτά τα όπλα. Επίσης υπάρχει συμφωνία για τη μη ανάληψη δράσης πόντισης Θα ήθελα να τονίσω πως το ζήτημα των χημικών όπλων δεν είναι καινούριο στην Ευρωπαϊκή Ένωση συζητείται σε διάφορα θεσμικά όρθια Ευρωπαϊκής Ένωσης από διάφορες οπτικές γωνίες, περιλαμβάνουμε το περιβάλλον, την ασφάλεια και τις επιπτώσεις. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στην απόφαση 285.0 του 2000 έθεσε ένα κοινοτικό πλαίσιο για την απαγόρευση αυτή της πώλησης ε, της ε, μεγαλύτερης συνεργασίας ώστε να μπορούν τα κράτη-μέλη να ανταποκριθούν στις ε, κατεπίγουσες καταστάσεις όπως για τις πετρελοκυλίδες κλπ. Η σύμβαση του Λονδίνου 1992 και το πρωτόκολλο του 1996 απαγορεύουν την διάθεση χημικών και βιολογικών παραγόντων στο πλαίσιο της Σύμβασης για την Προστασία της, ε, του θαλάσσιου περιβάλλοντος στην Σύμβαση ΟΣΠΑΡ που ετέθησε ισχύ το 1998 διάφορες πτυχές που ασχολούν, ασχολούνται με την πόντιση χημικών όπλων και πυρομαχικών τη Σύμβαση για τα Χημικά Όπλα που ετέθησε ισχύ το 1997 απαγορεύει την παραγωγή, την αγορά, την αποθήκευση, την μεταφορά και τη χρήση χημικών όπλων και απαιτεί την καταστροφή όλων των αποθηκευμένων χημικών όπλων. Η Σύμβαση για τα Χημικά Όπλα δεν καλύπτει την πόντιση χημικών όπλων πριν από το 1985. Εν τω μεταξύ η Σύμβαση αφήνει τα κράτη-μέλη τη δυνατότητα να αποφασίσουν να δηλώσουν κατά πόσο έχουν πωλήσει όπλα πριν από 1985. Η σύμβαση αναθέτει στα κράτη-μέλη να αποφασίζουν για την πόνηση των όπλων. Παρά το ότι η σύμβαση για τα χημικά όπλα δεν αφορά τα χημικά όπλα που ποντίστηκαν πριν το 1985, η ΟΑΧΟ μπορεί να χρησιμεύσει ως σημαντικό φόρουμ για την εθελούσια συνεργασία ανάμεσα στην οργάνωση αυτή, τα κράτη-μέλη, την ε, τεχνική γραμματεία και άλλες οργανώσεις που ασχολούνται με το ζήτημα της πόνης χημικών απλών. Μετά από την ε, δεύτερη αναθεώρηση της ε, σύμβασης, η Λιθουανία έχει ανλάβει διάφορες δραστηριότητες για μια καλύτερη διεθνή συνεργασία σχετικά με την πόντιση χημικών όπλων. Η Λιθουανία έχει, έχει θέσει το ζήτημα στην Ηνωμένα Έθνη και έχει αναλάβει πολλές διμερείς πρωτοβουλίες. Η Λιθουανία επιθυμεί η εσελούσια συνεργασία ανάμεσα στα κράτη-μέλη και ανάμεσα στις διεθνείς οργανώσεις με την βοήθεια της Ευρωπαϊκής Ένωσης θα οδηγήσουν σε μια αναθεώρηση των μητρώων για να εντοπιστούν πιθανοί χώροι για την πόντιση χημικών όπλων και πυρομαχικών. να υπάρξει ενημέρωση σχετικά με το που έχουν πονηστεί χημικά όπλα να συνεχιστούν οι δραστηριότητες για να ενημερωθεί το κοινό για ενδεχόμενους κινδύνους που μπορούν να προέλθουν από τα ποντισμένα στη θάλασσα χημικά όπλα και να εντοπίσει κατάλληλες δράσεις για να μετριάσει αυτόν τον κίνδυνο. Τέλος, να αναπτύξει τις ε, δραστηριότητες ενημέρωσης και την εξέβρεση υλικών που θα μπορούσαν να βοηθήσουν στην ε, μεγαλύτερη ασφάλεια. Και τέλος, θα πρέπει να υπάρξει μια ευρύτερη συνεργασία στην, ανάμεσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση και άλλες οργανώσεις. Στην... Διότι μόνο έτσι θα μπορέσουμε να περιορίσουμε τους κινδύνους που ενδέχεται να προκύψουν από την πόνηση και ευχαριστώ Πρόεδρε να πω ότι το κείμενο των παρατηρήσεών μου και ένα, ένα non-paper της Λιθουανίας είναι έγγραφα τα οποία έχω υποβάλει μαζί με ένα CD από το σεμινάριο που είχαμε οργανώσει στο Βίλνιους πέρυσι. Και υπάρχει και δήλωσή μου στα Ηνωμένα Έθνη από το 2008. Ευχαριστώ και αν υπάρχουν ερωτήσεις σχετικά με τη θέση μας, ευχαρίστω να σας απαντήσω. Μικρόφωνο παρακαλώ. Ο πρόεδρος μιλάει εκτός μικροφώνου. Α, Εντάξει. Λοιπόν, ναι, ήταν εκτός μικροφώνου ο πρόεδρος. Ε, σας ευχαριστώ πάρα πολύ και μας ενδιαφέρουν ιδιαίτερα τα στοιχεία του κόστους. Ε, τι κόστος επιφέρει, επιφέρουν όλες αυτές οι ενέργειες και αν υπάρχει δυνατότητα ανακύκλωσης αυτών των υλικών από τη στιγμή που ανακτώνται από τον πισμένα της θάλασσας. Με τα απαραίτητα επίπεδα ασφαλείας βεβαίως. Ε, έχουμε τώρα λίγο χρόνο στη διάθεσή μας για συζήτηση και δίνω το λόγο στον κύριο Λαντσμπέργκης. Ευχαριστώ. Με ενδιαφέρει πολύ το θέμα αυτό βέβαια και χαίρομαι που μας δόθηκε ευκαιρία για αυτή τη συζήτηση εδώ. Παρόλο που ε, δεν φτάνει διόλου ο χρόνος που έχουμε στη διάθεσή μας είναι ανεπαρκέστατος θα πρέπει να κάνουμε μια ενδελεχή συζήτηση για όσο χρόνο χρειάζεται να συζητήσουμε τα θέματα και να επιστήσουμε την προσοχή του σώματος και όλης της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε αυτό το ζήτημα. Διότι, όπως αντιλαμβάνεστε, όλα αυτά αντιπροσωπεύουν ένα τεράστιο κίνδυνο στα, κράτη, στα παράκτια κράτη της Βαλτικής. Και υπάρχουν εκατομμύρια άνθρωποι που θέλουν να ζήσουν στις περιοχές αυτές και δεν θέλουν να ε, ζήσουν σε μια ε, μολυσμένη περιοχή, σε μολυσμένα παράλια γνωρίζοντας ότι τεράστιες ποσότητες ε, όπλων έχουν ποντιστεί στη, στο, στη θάλασσα. Πιστεύω ότι πρέπει αυτή τη στιγμή να ε, κάνω μία ερώτηση και αργότερα όταν θα βρούμε τον κατάλληλο χρόνο θα κάνω τις γενικές μου παρατηρήσεις. Ήθελα λοιπόν να ρωτήσω μετά από αυτά που άκουσα τι γίνεται με την έλλειψη πληροφοριών που έχουμε, πληροφόρηση για τις ε, τοποθεσίες εκείνες όπου έχει γίνει dumping. Από ό,τι άκουσα ε, από τον κύριο Κόχ ανέφερε τις περιοχές του Σκάγερακ. Ε, στη, στη δική μας ε, μεγάλη περιφέρεια της Βαλτικής θάλασσας αντιμετωπίσαμε συγκεκριμένες ιστορικές πραγματικότητες όπως ξέρετε και η Βαλτική Συνέλευση, στην οποία ε, έχω εργαστεί, ε, Έχω μελετήσει αυτό το θέμα από το, την περίοδο 2000-2002 και ε, καταφέραμε να φτιάξουμε μια γενική εικόνα της κατάστασης. Από ό,τι θυμάμαι, Η απόφαση για το ντάμπινγκ αυτών των όπλων έγινε από τους νικητές του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου και έγινε το ντάμπινγκ αυτό σε διαφορετικές περιοχές της Βαλτικής αλλά έγινε και στον Ατλαντικό αρχικά. Εν συνεχεία το ντάμπινγκ δεν συνεχίστηκε στον Ατλαντικό, αλλά συνεχίστηκε στη Βαλτική. Μεταφέρθηκε δηλαδή στη Βαλτική, στην Ανατολική μάλιστα Βαλτική, περιοχή της Βαλτικής, η οποία ήταν ένα πολύ πρόσφορο, μια πρόσφορη τοποθεσία για το Σοβιετικό στρατό. από τους δυτικούς συμμάχους τώρα το dumping έγινε ε, υπό τη μορφή του φορτίου αυτού πάνω σε πλοία. Οι Σοβιετικοί δεν εφάρμοσαν αυτή την, το αίτημα των δυτικών να φορτωθεί ε, να φορτωθούν αυτά τα απόπειτα σε πλοία και συνεχεία να ποντιστούν, αλλά έκαναν μία διάχυση, μία διασπορά της αναπόθεσης ε, των ε, αποβλήτων αυτών σε διάφορες περιοχές τις οποίες δεν ξέρουμε. Και αυτό βεβαίως ε, είναι ένας κίνδυνος, μεγάλος κίνδυνος σήμερα. Παρόλο που υπάρχει αυτή η κατάσταση δεν, μας, δεν επιτρέπεται να μην συνεχίζουμε τις προσπάθειές μας σήμερα και να, να εργαστούμε πάνω σε αυτό το θέμα, να μελετήσουμε αυτό το θέμα. πρέπει βεβαίως να βασίσουμε όλες μας τις εργασίες μας σε συγκεκριμένα στοιχεία. Όταν παρεμβαίνει ιστορία και όταν μιλάμε για λιμένες αποφάσεις, τα πράγματα δυσκολεύουν. Διότι, όπως είπα, έχουμε χίδιν, χίδιν απόρριψη όπλων, ενό οπλοστασίου από εδώ και από εκεί, αλλά έχουμε και οργανωμένη ε, πόντιση πάνω σε πλοία, από πλοία. Επειδή λοιπόν έχουμε τις δύο αυτές διαφορετικές μορφές ε, πόντισης, πολλά, ορισμένα κράτη-μέλη μπορεί να μην θέλουν να εμφανίσουν τις πληροφορίες αυτές. Όμως θα πρέπει στα αρχεία των κρατών αυτών να υπάρχουν πληροφορίες τις οποίες να μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε. Πιστεύω ότι θα, πρέπει να έχουν καταγραφεί τα στοιχεία αυτά σε παλιά αρχεία. Και εάν δεν μπορέσουμε να εντοπίσουμε τις τοποθεσίες αυτές θα αντιμετωπίσουμε έναν μεγάλο κίνδυνο. Γι' αυτό θα πρέπει να προβάλλουμε αυτό το πρόβλημα και να μην ε, θέλουμε να αποφύγουμε και τις πολιτικές διαστάσεις. Υπάρχουν οπωσδήποτε πολιτικές διαστάσεις σε αυτό το επικίνδυνο γεγονός. Ε, θέλετε να αντιμετωπίσουμε στο μέλλον μια τεράστια καταστροφή Εάν αυτές οι πληροφορίες που σίγουρα υπάρχουν σε κρατικά αρχεία παραμείνουν μυστικές, πιστεύω ότι αυτή η μυστικότητα αγγίζει τα όρια της, ε, του εγκλήματος. Είναι εγκληματική, διότι θα οδηγήσει αναπόφευκτα σε μια τεράστια καταστροφή. Και πάλι, λοιπόν, το πρόβλημα δεν είναι επειδή δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι να μην κάνουμε τίποτα. Αυτή τη στιγμή περιμένουμε. Είμαστε σε στάση αναμονής. Η στάση αυτή αναμονής είναι ανεύθυνη. Λείπει η υπευθυνότητα. Η ιδέα της κατασκευής σαρκοφάγων ε, εκεί όπου ε, εντοπίζονται πλοία που έχουν τέτοια χημικά είναι μία ιδέα, αλλά ε, τι θα κάνουμε, γιατί εκεί ξέρουμε, μπορούμε να εντοπίσουμε τη χωματερή, την, την, την πόντιση που έγινε. Τι θα γίνει όμως με την χίδη πόντιση ε, όπλων, ε, χημικών όπλων, όπου δεν μπορούμε να τα εντοπίσουμε συγκεντρωμένα κάπου. Νομίζω ότι θα πρέπει να γίνει μία έκθεση η οποία να προωθηθεί σε ένα υψηλό διεθνές επίπεδο για να ε, ασκηθεί πίεση στην ε, δημοσίευση των μυστικών αυτών αρχείων που ε, θα βοηθήσουν στον εντοπισμό των ποντισμένων χημικών, διότι αυτή η μυστικότητα είναι, όπως είπα, ανεύθυνη και επικίνδυνη. Εάν λοιπόν ανακτηθούν αυτά τα χημικά όπλα τα οποία καλύπτουν μία τα οποία καλύπτουν όλες τις πτυχές ε, της ε, Σύμβασης για την Απαγόρευση Χημικών Όπλων υπάρχει σαφώς ενδιαφέρον από διάφορα κράτη να μην ανακτηθούν να μην ανακτηθούν και αποκαλυφθεί το μέγεθος του κινδύνου. Όμως ε, καταλαβαίνετε ότι εδώ επισέρχονται και εμπορικά κριτήρια διότι έχουμε την κατασκευή του, των αγωγών και στην κατασκευή των αγωγών εμπλέκονται διάφορες εταιρείες οι οποίες μπορούν να ασκούν ε, πιέσεις Πιστεύω ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θα πρέπει να εκδώσει ένα ψήφισμα ε, και να ζητήσει με έντονο τρόπο την ανάληψη δράσης. Μέχρι τώρα όμως όλα αυτά έχουν αραχνιάσει. Ας πούμε, ζητούμε την διεξαγωγή ερευνών. Εάν όμως η Gazprom πληρώνει τους ερευνητές να ε, συντάξουν μία έκθεση και η Gazprom είναι αυτή που έχει τα μεγάλα συμφέροντα για την κατασκευή του αγωγού τότε ε, ε, επισερχόμεσα σε ακόμα πιο επικίνδυνα πεδία παραδείγματος χάρη του καουμπόικου καπιταλισμού από πλευράς Ρωσίας που δημιουργεί μεγάλους κινδύνους για τα άλλα κράτη. Θα ήθελα λοιπόν να ακούσω από τους εισηγητές τι βήματα μπορούν να αναλυφθούν από ένα πολιτικό σώμα όπως είμαστε εμείς. For the very interesting uh, questions you but we, we need some time for... Κοιτάξτε, χρειαζόμαστε και λίγο χρόνο για τις απαντήσεις, ενδιαφέρουσες ερωτήσεις, αλλά πρέπει να έχουμε χρόνο και για τις απαντήσεις. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ε, εδώ και πολλά χρόνια υπάρχει ε, μια διαμάχη για το κατά πόσον αυτές είναι ορολογιακές βόμβες οι οποίες έχουν ποντιστεί στη θάλασσα, ε, πότε θα εκραγούν ή μήπως είναι καλύτερα ε, να συνεχίσουν να σκουριάζουν στον πυθμένα της θάλασσας. Ευχαριστώ πολύ για τις πληροφορίες. Εδώ και πολλά χρόνια ε, προσπαθώ να βρω ποιος φέρει την πολιτική ευθύνη. Θα είμαι σύντομη. Στη Βόρειο Γερμανία ε, στο Schleswig Holstein, ρώτησα στο κρατήδιο αυτό ε, στο βορρά της Γερμανίας, πού είναι το μητρό όπου αναφέρονται αυτά τα κατάλοιπα. Μου είπαν δεν υπάρχει τέτοιου είδου ε, μητρό, τα ρώτησα στο Αμβούργο. Πού βρίσκεται τέλος πάντων αυτό το, αυτός ο κατάλογος με εγκαταλειμμένα πυρομαχικά γιατί σε τελική ανάλυση δεν είναι μόνο ε, πυρομαχικά αλλά είναι και φόσφορος ε, και άλλα έτσι συμπαθή προϊόντα που εγκαταλείφθηκαν εκεί. Και στο Αμβούργο δεν μου είπανε τίποτα. Έτσι λοιπόν ως πολιτικός εγώ προτιμώ να έχω μια φιλελεύθερη ε, συντηρητική κυβέρνηση ε, γιατί εκεί μπορώ να ασκήσω πίεση. Ε, μου είπανε βέβαια ότι το Υπουργείο Περιβάλλοντος δεν είναι αρμόδιο, το Αμήνης δεν μπορεί να δώσει πληροφορίες και τελικά η κυβέρνηση της Γερμανίας είπε ότι το τι συνέβη σε εποχές ε, Ανατολικής Γερμανίας έτσι και αλλιώς δεν είναι αρμοδιότητα της Ενωμένης Γερμανίας. Ως εκ τούτου <clears throat> δεν έχουν ιδέα που βυθίστηκε τι. Γιατί και η Γερμανία ε, μετά την ήττα στο Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο πόντισε πυρομαχικά στη θάλασσα. Ακόμα και η δημοτική ε, αυτοδιοίκηση δεν θέλει να αναφέρει που υπάρχουν διαπυρομαχικά και στις ακτές. Άνθρωποι τραυματίστηκαν. Ε, ψαράδες, ε, αν ψαρέψουν ε, πυρομαχικά αμείβονται. Αυτό όμως είναι παράλογο γιατί οι ψαράδες δεν είναι εκπαιδευμένοι για να συλλέγουν πυρομαχικά. Ως εκ τούτου καταργήθηκε και αυτή η διάταξη. Μίλησα με τους ψαράδες και με πλειοκτήτες και μου είπανε επειδή δεν πληρωνόμαθε πιάνουμε τις βόμβες και τις ξαναπετάμε μέσα στη θάλασσα. Και τι κάνουν δηλαδή, τις παίρνουν δεξιά-αριστερά, δεν τις πετάνε αμέσω μέσα, τις πάνε πιο εκεί και τις πετάνε παρακάτω τη νύχτα α πούμε για να μην τους βλέπουν. Τώρα, όσον αφορά την ε, πολιτική ευθύνη, τη συζητήσαμε αυτή στην ε, Πράσινη Βίβλο και νομίζω ότι κατατέθηκαν πολύ καλές προτάσεις για τη συνεργασία. Εγώ μόνο που έχω την εντύπωση ότι λείπει η πολιτική βούληση ε, και πρέπει να αναζητήσουμε και την ε, διάθεση χρηματοδότησης. Δηλαδή όπου υπάρχουν αυτά τα πολεμαχικά να εξεταστούν ποια είναι η κατάστασή τους, πόσο κοστίζει. Τώρα το κάνουμε ας πούμε στον ε, αγωγό γιατί να γίνεται και εκεί να μην γίνεται αλλού. Και να πω και κάτι άλλο που είναι το πρόβλημά μας. Όπως και με τις ε, νάρκες που έχουν ποντιστεί στη γη όταν λιώνει το χιόνι, κάθε χρόνο στέλνουμε στο του παραδείγματος χάνει ε, ειδικού που ψάχνουν ε, να βρουν ε, τις νάρκες για να μην εκραγεί καμία. Ίσως βέβαια οι νάρκες αυτές δεν είναι λίγο πιο πέρα και εκεί πια πάβουν να ψάχνουν. Τα λέω αυτά για να σας πω, εντάξει δεν θέλω να σπείρω τον πανικό, αλλά πρέπει να βρούμε τη δυνατότητα μέσα από τα Εθνικά Κοινοβούλια και σε συνεργασία με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Δεν προχωράω τόσο εσείς να βρούμε τους υπέτειους, γιατί αν το κάνουμε αυτό δεν θα προχωρήσουμε ποτέ. Τον κίνδυνο πρέπει να ελέγξουμε. Ως εκ τούτου πρέπει να υπάρχει ε, συντονισμένη συνεργασία στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Και νομίζω αυτό ε, κατέστη απόλυτα σαφές την περασμένη εβδομάδα στις ακτές της Νορβηγίας ε, είναι ένα μέτρο το οποίο αφορά όχι μόνο τη δική μας την υποπιτροπή, θα πρέπει τις ε, πληροφορίες να τις δώσουμε περαιτέρω ε, στην Επιτροπή Ελίας και σε άλλους και να προσπαθήσουμε σε επίπεδο κυβερνήσεων να ασκήσουμε πίεση για να αναλυφθούν ευθύνε ε, για τους ανθρώπους αλλά και για το περιβάλλον. Και δεν αρκεί απλά να σημαίνει αυτό που γίνεται τώρα στη Γερμανία με το να δοκιμάζει κανείς νέες τεχνολογίες με την αφαίρεση πάνω οξυγόνου γιατί ο κίνδυνος υπάρχει είναι όπως τα ε, πυρομαχικά θα κραγούν και θα πεταχτούν και στον αέρα όλοι οι ψαράδες που ψαρεύουν. Θεωρώ λοιπόν ότι πρέπει να εξετάσουμε πολύ προσεκτικά το όλο θέμα και να διευκρινιστεί επίσης το θέμα της πολιτικής ευθύνης. Ε, πολύ ωραία, δεν ξέρω τώρα, ε, θα απαντήσετε βέβαια, αλλά αν έχετε την καλοσύνη να είστε πολύ σύντομοι, ε, γιατί δεν έχουμε χρόνο. Ε, το πρόβλημα είναι πολύ σημαντικό, αλλά λυπάμαι πάρα πολύ. Δυστυχώς πέσαμε σε πίεση χρόνου. Και θα δώσω πρώτα το λόγο στον κύριο Χάρτ. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ για τα σχόλια. Ήταν πολύ πετυχημένα. Θα ήθελα να δώσω μερικέ σύντομε απαντήσει ε, σε όσες περισσότερες ερωτήσεις γίνεται. Τώρα σχετικά με την τεχνική εφικτότητα θα πρέπει να πετύχουμε το σωστό μείγμα ε, νομικών εμπειρογνωμόνων, τεχνικών ε, επιστημών κλπ. Πάντως είναι δύσκολο να απαντήσει κανείς ε, ναι ή όχι αν είναι εφικτό από τεχνική σκοπιά ε, για την ανάκτηση των πυρομαχικών σε μερικές περιπτώσεις, ναι. Υπάρχουν κάποιες ε, διαδικασίες για την αναζήτηση πυρομαχικών όπου υπάρχουν δίτες και λοιπά εκπαιδευμένοι. Δεν υπάρχει μια εύκολη απάντηση ναι ή όχι. από τις λεπτομέρειες τώρα σε ό,τι φορά το κόστος είναι δυνατόν σε τέτοιες περιπτώσει να κάνουμε εκτίμηση του κόστους ένα είδος εκτίμηση είναι αυτή που γίνεται με βάση πολιτική δέσμευση όπου αποφασίζεται να δαπανηθούν ορισμένα χρήματα σε, για κάποιες και ένα τρόπος είναι ε, ο τρόπος bottom-up. Όταν ακολουθήσετε αυτή την μέθοδο, μία από τι αβεβαιότητες είναι πως ε, διαδικασία για την... Υπάρχει μια διαδικασία για την εξέβρεση τεχνικών ε, δυνατοτήτων. Αλλά πολλές φορές αυτό δεν μπορεί να γίνει δεκτό από πολιτική σκοπιά, γιατί μπορεί να υπάρξει, υπάρχουν απώλειες ζωής. Ίσως ο κ. Κότσου να μπορούσε να μας πει πώς ε, το γερμανικό πρόγραμμα διάθεσης ε, πυρομαχικών ήταν αποτελεσματικό, αλλά μια να για αναφορά στο αμερικανικό πρόγραμμα υπάρχουν ε, κάποιοι χώροι που είναι διαθέσιμοι. Ένα αυτό είναι το Mr. Facility που ασχολείται και με χημικά αλλά και με συμβατικά όπλα και Στην παρουσίασή μου δεν είπα πολλά πράγματα σχετικά με το θέμα αυτό, αλλά προσπάθησα να παραμείνω μέσα στα χρονικά όρια. Με αυτό είναι δικό μου πρόβλημα. Συμφωνώ και ενδιαφέρομαι ιδιαίτερα με την ιστορική πτυχή. Μπορείτε να δείτε πολλές λεπτομέρειες Υπάρχουν προφορίες για την ε, Μαύρη Θάλασσα, την Μεσόγειο αλλά και τη Βαλτική. Κατά την άποψή μου, η Μεσόγειος ε, και η Μαύρη Θάλασσα προσφέρουν ενδιαφέρον διότι εκεί έχουν ποντιστεί σημαντικές ποσότητες ε, όπλων και πυρομαχικών. Έγιναν σχόλια σχετικά με την πολιτική διάσταση ναι, είναι δυνατόν να γίνει πολιτική ανάλυση, αλλά όπως προείπα, εμείς ετοιμάσαμε ένα έγγραφο ενημερωτικό, μπορεί να κάνουμε πούμε, σε μια σε βάθος ανάλυση. Νομίζω ότι το ζήτημα των, του αγωγού έχει εξεταστεί από σημαντικές ε, μελετητικές εταιρείες. Εμείς ε, σεβόμαστε τα ευρήματά τους και αυτό το οποίο έκανε αυτή είναι προσωπική μου άποψη φυσικά. Θα γίνουν ευμενώς αποδεκτά, τα, οι θα διανεμηθούν. Τώρα, έχουν, δεν έχουμε μόνο τα τεχνικά στοιχεία, αλλά έχουμε και τα πολιτικά αυτό μπορεί να είναι μια άλλη ιστορία, αλλά πολιτικές, αλλά σίγουρα θα υπάρχουν πολιτικές θεωρήσεις. αλλά κάτι να προχωρήσω. Κάτι ακόμα. Στο τέλος αναφέρθηκε το θέμα της έλλειψης ενημέρωσης σχετικά με τις τοποθεσίες ε, στις ε, ακτές της Γερμανίας. Υπάρχουν κάποιες προφορίες διαθέσιμες, αλλά εξαρτάται το πώς προσεγγίζει κανείς ε, την αναζήτηση πληροφορίας. Υποθέτω πως με τα όσα μας είπε ο κύριος Κότς, πολλά από αυτά θα μπορούσαν να αναζητηθούν. Δεν θα ήθελα να σχολιάσω πολλά από τα άλλα που υπόθηκαν για την ευρωπαϊκή πολιτική, τι θα πρέπει να κάνει το Κοινοβούλιο. Θα ήθελα να απέχω από τέτοιου είδου παρατηρήσεις. Ο κύριος Σόσμπορν έχει το λόγο. Thank you, sir. Um, as όπως αναφέρθηκε και προηγουμένως, ε, προφανώς ε, σε μεγάλο βαθμό πρόκειται για πολιτικά θέματα. Εγώ είμαι τεχνικός, ε, κύριε, και μακράνε μου η πολιτική όσον αφορά ε, την απαγόρευση χημικών ε, όπλων, εμείς δεν μπορούμε να κάνουμε σχόλιο. Σε καθαρά τεχνικό επίπεδο θα ήθελα να επισημάνω ότι όσον αφορά την ανάκτηση των χημικών όπλων που βρίσκονται στο βυθμό της θάλασσας, ε, προηγούνται Πρωτοπόροι είναι οι Ιάπωνες και πολλά από αυτά που μάθαμε ε, τα μάθαμε παρατηρώντας τις δικές τους τις επιχειρήσεις. Ε, παράλληλα οι επιχειρήσεις αυτές είναι πολύ περιορισμένες. Σε περίπου τέσσερα χρόνια έχουν ανακτήσει και καταστρέψει περίπου 3.000 χημικά όπλα. Βέβαια σε όλες αυτές τις περιπτώσεις ε, σε βάθος περίπου 10 μέτρων με πολλές δυσκολίες η καταστροφή αυτών των όπλων είναι εφικτή. Υπάρχει τεχνολογία. Ε, αυτή τη στιγμή η τεχνολογία υπάρχει στην Ιαπωνία, στην Κίνα, στη Γερμανία και μπορεί και να μεταφερθεί. Είναι λοιπόν δυνατή η καταστροφή. Όμως η ανάκτηση είναι το δύσκολο θέμα. Εκεί που αρχίζουν το τεχνικής φύσεως θέμα και εκεί υπάρχουν οι περισσότερες δυσκολίες. Παραδείγματο χάρη, ο εντοπισμός ε, αυτών των ε, όπλων, αυτά είναι καλυμμένα από άμμο και όταν ε, χρησιμοποιεί κανείς το μαγνήτη εντοπίζεται και πολλά άλλα στοιχεία μαζί με τα όπλα. Οι Ιαπωνέζες με για κάθε πυρομαχικό ε, τραβάνε με το μαγνήτη και χιλιάδες μέταλλα. Αυτό είναι πολύ δύσκολο και δημιουργεί πρόβλημα. Οι προλαλήσαντες, οι συνομιλητές ε, έκαναν κάποια σχόλια. Είναι λοιπόν σαφές ότι δεν έχει ε, καταστεί ε, σαφές το πρόβλημα. Όταν λαμβάνετε απόφαση για ανάκτηση όχι θα πρέπει να λαμβάνετε με βάση υγιείς πληροφορίες. Και όπως αναφέρθηκε ήδη, ε, μερικοί πρέπει να εστιάσουν την προσοχή τους σε αυτό το θέμα. Κοιτάξτε, ε, λυπάμαι, αλλά άλλα τέσσερα λεπτά έχουμε για ταυτόχρονη διερμηνία. Αν έχει την καλοσύνη ε, να το λάβετε υπόψη σας, γιατί εγώ θα ήθελα να δώσω το λόγο και στον κύριο πρέσβη. Μία παρατήρηση μόνο από μένα τεχνικής φύσεως. Στην Ιαπωνία είχαμε ένα project όπου ανακτήσαμε χιλιάδες χημικά όπλα από, με δίτες Αυτή τη στιγμή βεβαίως δεν θέλουμε να έχουμε δίτες που κάνουν αυτό το επικίνδυνο έργο θέλουμε να χρησιμοποιήσουμε τη ρομποτική έτσι ώστε να μην χρησιμοποιούμε δίτες επιτόπου από την άλλη πλευρά άλλη, μία πολύ καλή αντιμετώπιση της ε, τεχνικής ας πούμε ορατότητας είναι το water cutting water cutting σημαίνει ότι κόβουμε, τεμαχίζουμε τα συμβατικά όπλα σε κομμάτια και εν συνεχεία τα μεταφέρουμε τεμαχισμένα στην εγκατάσταση καταστροφής. Δύο λοιπόν, πρα, δύο λοιπόν ε, εργαλεία αν θέλετε θα παρουσιαστούν στην αγορά ε, σε δύο-τρία χρόνια. Το water cutting, ο τεμαχισμός υπό το νερό δηλαδή, τεμαχισμός των ε, αντικειμένων αυτών, όπλων αυτών, κάνουμε πειράματα αυτή τη στιγμή στη Γερμανία και η ρομποτική. Ε, επίσης στα, στην Αλία, εδώ το θέμα είναι, το ζήτημα είναι πολύ σημαντικό. Important lobby maybe. Um, we had uh, these numbers of incidents uh, in the Danish fishery talking of 450 incidents ah, ναι. incidents uh, concerning the Danish fishery. Άρα, και τα, τα, οι αριθμοί αυτοί έχουν αυξηθεί κατά 20 ή 30 όταν καταβλήθηκαν αποζημιώσεις για τον, ε, την απώλεια αλλιευμάτων. Καταλαβαίνετε ότι στην ε, αλία η επιβίωση των ψαράδων εξαρτάται από τα αλλιεύματα που πιάνουν και βεβαίως έγιναν ε, ε, προτάσεις να απογορευτεί η αλία σε συγκεκριμένες επικίνδυνες περιοχές λοιπόν τα οποία αυτή τη στιγμή συμβαίνουν δεν, δεν μπορούμε να τα, δεν, δεν ξέρουμε, δεν τα έχουμε καταγράψει δηλαδή πόσα επικίν, πόσες επικίνδυνες ουσίες βγαίνουν προσωρινά ή ψαρεύονται από τη θάλασσα και εν συνεχεία και πάλι από τους ψαράδες για να τα ξεφορτωθούν. Ο κύριος ε, Πρέσβης έχει ακόμα δύο λεπτά πριν τελειώσουμε. Ευχαριστώ. Θα είμαι τηλεγραφικός. Ε, ε, εγώ κατά κάποιο τρόπο αντιπροσωπεύω την πολιτική πλευρά. Ό, όλοι οι προλαλήσεντες είναι επιστήμονες. Θα ήθελα λοιπόν να τονίσω ότι η Λιθουανία ε, εδώ και δύο χρόνια ενθαρρύνει τα κράτη-μέλη που έχουν συνυπογράψει τον ΟΑΧΟ, τον οργανισμό αυτό, να συζητηθεί το θέμα της πόντισης, της, του ντάμπινγκ χημικών όπλων ο βασικός μας στόχος. Δεν είναι ούτε να τροποποιήσουμε ούτε να αλλάξουμε την συνθήκη για τα χημικά όπλα, αλλά να επιστήσουμε όσο το δυνατόν περισσότερη προσοχή ε, στο πρόβλημα αυτό, ώστε να το σημειώσουν όλες οι χώρες ε, και οι διεθνείς οργανισμοί, να το λάβουν σοβαρά υπόψη τους. Γι' αυτό ενθαρρύνουμε τη συζήτηση και επίσης ενθαρρύνουμε τη συζήτηση αυτή για να προετοιμαστεί ένα γόνιμο έδαφος πολιτικής συζήτησης. Ε, ανεξάρτητα από το τι τεχνικές λύσεις θα βρεθούν στο ενδιαμέσως. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ όλους τους, τους συμμετασχόντες σε αυτή την ακρόαση. Οι κίνδυνοι είναι σαφείς, έχουν καταγραφεί. Πρέπει να καταλήξουμε συμπεράσματα και να συντάξουμε ένα κατάλογο προτεραιοτήτων η επόμενη μας ενέργεια είναι να αποφασίσουμε ακριβώς ποιες είναι προτεραιότητες. Ο αγωγός ε, είναι εξωτερικό στοιχείο, ο αγωγός ε, πετρελαίου φυσικού αερίου, ε, αλλά το πρόβλημα παραμένει. Σας ευχαριστώ πολύ γιατί με τις ενέργειές σας προσπαθείτε να προστατεύσετε και την αλή και τις παράκτιες περιοχές. Το επόμενο βήμα είναι στα χέρια μας και αυτό πρέπει να αποφασίσουμε ποιο θα είναι. Ευχαριστώ πολύ.